Καλημέρα σας, μια ωραία καλημέρα σε όλους. Εδώ, στο τροπικό κλίμα της αίθουσα συνεδριάσεων. Σε αντίθεση με την παγωνιά έξω, εδώ βράζει η αίθουσα. Λοιπόν, πρώτον, έγκριση της ημερήσιας διάταξης <coughs> μπορεί να εγκριθεί, φαντάζομαι, όσο έχει. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ή επιθυμίες για αλλαγές. Δεύτερον, ανακοινώσει του Προέδρου. Έχουμε όλες τις γλώσσες σήμερα, με εξαίρεση τα μαλτεζικά, τα κροατικά και τα γοεζελικά. Και αύριο ε, θα έχουμε μαλτέζικα και τις άλλες δύο όχι. Έχουμε και ένα νέο μέλος στην Επιτροπή μας, μετά την παρέτηση της Ινές Ζούμπερ από την ε, Ενωτική Αριστερά. Ήρθε ο κύριος Ζωάου Πιμέντα Λόπες, τον οποίο και καλωσορίζουμε θερμά ή θα τον καλωσορίσουμε όταν έρθει, διότι αυτή τη στιγμή ακόμα απουσιάζει. Τρίτον, έχουμε επισκέπτες 30 από την ε, περιοχή Λιμουζάν που ατού Σαράν, τη Γαλλία, ε, που έχει καλέσει η κυρία Μωρέν Σατιέ, 10.30 με 11.30 θα έρθουν και 11 μέλη του Νορβηγικού Κοινοβουλίου. Αυτοί είναι οι επισκέπτες μας που θα μας έρθουν στις 18 του μηνός, αύριο δηλαδή 9 με 11.30. Έγκριση των πρακτικών τρίτο θέμα των συνεδριάσεων στις 12 και 13 Οκτωβρίου και 26 Νοεμβρίου 2015. Αν δεν έχετε σχόλια και παρατηρήσεις θα θεωρηθούν τα πρακτικά εγκεκριμένα. Πάμε λοιπόν στο σημείο 4 έκθεση σχετικά με την εφαρμογή τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία με ιδιαίτερη έμφαση στις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής CPRD του ΟΗΕ. Είναι πολύ μακρύς ο τίτλος. Καλωσορίζω όλους τους ε, ενδιαφερομένους και τους συμμετέχοντες πριν μπούμε στη συζήτηση. Μια σύντομη παρατήρηση. Έχουμε νοηματική γλώσσα, διερμηνία και θα βρείτε τρεις κάρτες. Η πράσινη είναι ότι έχετε καταλάβει ε, και είναι όλα καλά. Η κίτρινη κάρτα σημαίνει, ε, βγάζω κίτρινη κάρτα στον ομιλητή γιατί μιλάει πάρα πολύ γρήγορα. Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Γιατί οι διερμηνείς δεν σας προβαίνουν όχι μόνο της νοηματικής και οι δικοί μας συνάδελφοι στις καμπίνες έχουν τεράστιες δυσκολίες όταν μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα και η κόκκινη κάρτα σημαίνει δεν κατάλαβα τίποτα. Παρακαλώ επαναλάβετε τα όσα είπατε με πιο απλά λόγια για να τα καταλάβω. Ελπίζω να τα είπα σωστά αυτές τις τρεις κάρτες που είναι σαν φανάρι και με αυτό το σύστημα μπορούμε να προχωρήσουμε. Αν κάποιο πάρει κόκκινη κάρτα δεν πρέπει να φύγει για τα ποδητήρια όπως είναι, μπορεί να παραμείνει στην αίθουσα. Εντάξει, λοιπόν, σας Καλωσορίζω και τους προσκεκλημένους του Diane Kingston από την Επιτροπή αυτή του ΟΗΕ και επίσης παρευρίσκεται ο κύριος Μάικλ Φλάχερτη που είναι Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επίσης καλωσορίζω την Έμιλη Οράιλι που είναι η διαμεσολαβήτρια, όχι η διαμεσολαβητής του Κοινοβουλίου, έτσι, λέγοντα αυτά τα πράγματα και Γιούντα Άνκα που είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αναπηρίας και επίσης το Γιάν Γιάραπ, που είναι ο περιφερειακός εκπρόσωπος της ΥΠΑ της Αρμοστίας του για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτοί είναι προσκεκλημένοι, τους καλωσορίσαμε και τους πέντε εμπειρογνώμονες που θα μιλήσουν στον πρώτο γύρο 10 λεπτά ο καθένας. Ξέξα κανέναν. Diane Kingston, σας είπα πρώτη. Πρώτη πρώτη σας ανέφερα. Πέντε εμπειρογνώμονες λοιπόν, δέκα λεπτά έκαστος και θα ακολουθήσουν οι εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές της Επιτροπής Απασχόλησης. Η κυρία Κίνγκστον λοιπόν έχει πρώτη το λόγο. Παρακαλώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να έρθω εδώ να μιλήσω μαζί σας σήμερα μου ζητήθηκε να αναφερθώ σε διάφορα θέματα σχετικά με την αναθεώρηση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ε, Ατόμων με Αναπηρία. Αντί για CRPD θα αναφέρομαι στη Σύμβαση. Ε, θα μιλήσω για τον ρόλο της Επιτροπής σε την διαδικασία αναθεώρησης και κυρίως σε τις συστάσεις. Είμαι ένα από τα 18 μέλη της Επιτροπής της Σύμβασης. Ο ρόλος της Επιτροπής αυτής είναι να παρακολουθεί την εφαρμογή της σύμβασης. Αυτό γίνεται με μια περιοδική διαδικασία υποβολής εκθέσεων. Δύο χρόνια μετά την επικύρωση ή τη σύναψη στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλεται η αρχική έκθεση και μετά κάθε τέσσερα χρόνια υποβάλλεται έκθεση. Επίσης αναλαμβάνουμε και άλλες δραστηριότητε, αλλά αυτή είναι η πιο σημαντική από όσε θα μα απασχολήσουν σήμερα. Όσον αφορά την ε, διαδικασία αναθεώρησης, ε, ήταν ιστορική, διότι ήταν ε, ο πρώτος περιφερειακός φορέας που ασχολήθηκε με αυτό. Εξετάσαμε λοιπόν την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχαμε έναν κατάλογο ερωτήσεων ή θεμάτων που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο κατάλογος ερωτήσεων βασίστηκε σε όλες τις εκθέσεις, όχι μόνο των χωρών, αλλά και από μέλη της κοινωνίας των πολιτών και άλλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν είχε ένα διάστημα τριών μηνών για να απαντήσει στον κατάλογο των ερωτήσεων. και οι απαντήσεις αυτές σε συνδυασμό με τις ε, εκθέσεις ε, αποτέλεσαν τη βάση για τον εξάωρο διάλογο που πραγματοποιήθηκε στην Γενέβη. Από εκεί προέκυψαν 36 συστάσεις κλειδιά, εκ των οποίων οι τρεις ε, απαιτούσαν κάποια ε, συνέχεια εντός ενός τριμήνου, ενώ οι άλλες συστάσεις θα εφαρμοστούν μέσα στην επόμενη τετραετία μέχρι την επόμενη υποβολή έκθεσης. Θα επικεντρωθώ λοιπόν στις συστάσεις που αφορούν τους κύριους τομείς δεν γνώριζα πολύ καλά την Επιτροπή Απασχόληση. Ε, νόμιζα ότι ασχολείστε μόνο με την απασχόληση. Τώρα ε, διαπιστώνω ότι ασχολείστε και με άλλα θέματα. Η απασχόληση όμω είναι πολύ σημαντικό τομέα και θα ήθελα εδώ να τονίσω 11 ε, σημαντικού τομεί. Πρώτον, υπάρχουν πολύ υψηλά επίπεδα ανεργίας στα άτομα ε, με αναπηρίες, σε σύγκριση με τα άτομα χωρίς αναπηρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχουν ε, τα προστατευμένα εργαστήρια, συμμετέχουν κυρίως σε τέτοια και όχι στην ανοιχτή αγορά εργασίας, τα οποία χρηματοδοτούνται από κοινωνικές επιδοτήσεις κατόπιν ε, κοινωνική προστασία για τους ανθρώπους που δεν έχουν δουλειά και κυρίως μέτρα κοινωνικής προστασίας ε, που έχουν υποστεί περικοπές λόγω λιτότητας. Επίσης, ε, ελεύθερη κινητικότητα είναι ένας τομέας τον οποίο πρέπει να προσέξουμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα όσον αφορά την κινητικότητα ατόμων που χρειάζονται ειδική υποστήριξη κατά τις μετακινήσεις τους. Επίσης, ευαισθητοποίηση, κατάρτιση ε, στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα αναφερθώ λίγο στο ε, πλαίσιο παρακολούθησης που κατά τη γνώμη μου είναι προβληματικό εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η έλλειψη σημείων εστίασης. Επίσης, συντονισμός και συνεκτικότητα στις πολιτικές των διαφόρων θεσμικών οργάνων για να ε, μπορέσει να εφαρμοστεί πλήρως ε, αυτή η σύμβαση και για να μπορέσει ε, να φέρει αλλαγές στις ζωές των ανθρώπων με αναπηρίες θα πρέπει να γίνεται καλός συντονισμός στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός και μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Θα πρέπει να έχουμε όλη την ίδια παρτιτούρα, να το πω έτσι. Στα δεδομένα επίσης μπορείτε να αναλάβετε δράση, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξωτερικές δράσεις. Στις συστάσεις τονίσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μοναδική ευκαιρία να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή των ε, νέων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης ε, και του θεματολογίου για το 2030. Χρειαζόμαστε λοιπόν αναλυμένα δεδομένα, όχι μόνο αναφύλο και ηλικία, αλλά και ε, για τα άτομα με αναπηρίες. Και τέλος, και εξίσου σημαντικό, είναι η συμμετοχή ε, των ιδίων των ανθρώπων με αναπηρίες, ε, στα οποία θα αναφερθώ πιο αναλυτικά. Θα ήθελα λοιπόν να επικεντρωθώ σε, τέσσερις, σε τέσσερα σημεία του καταλόγου. Καταρχάς, άρθρο 33 μάλλον είναι το πιο παρεξηγημένο άρθρο της σύμβασης. Διαπιστώνω τώρα που ε, ε, έχω συμμετάσχει στον ε, διάλογο. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην εφαρμογή της σύμβασης και την παρακολούθηση της εφαρμογής. Και θα πρέπει αυτές οι δύο διαδικασίες να είναι τελείως ξεχωριστές η μία από την άλλη. Όσον αφορά την εφαρμογή, μίλησα για συντονισμό και συνεκτικότητα στις πολιτικές των διαφόρων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικροτώ το ότι η Επιτροπή της Σύμβασης ε, καλύπτει και τον συντονισμό. Η διαδικασία παρακολούθησης όμως θα πρέπει να είναι απολύτως ανεξάρτητη και αυτό το τόνισα στο πλαίσιο του επικοδομητικού διαλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί μέρος ε, του φορέα παρακολούθησης και επικροτούμε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα πια δεν συμμετέχει. Ωστόσο, Είναι επίσης σημαντικό η Επιτροπή απασχόληση η ΛΥΜΠΕ και η ΠΕΤΗ επίσης να μην συμμετέχουν στο πλαίσιο παρακολούθησης. Δεν μπορείτε να παίζετε και τους δύο ρόλους και να εφαρμόζετε και να παρακολουθείτε. Ε, ο έλεγχο ε, θα πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα. Για να είναι όμως αποτελεσματική η παρακολούθηση και για να υπάρχει συντονισμός ε, και συνεκτικότητα θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς πόροι. Για μένα ήταν κρίμα ότι τότε που το, ε, το focal point ήταν η Γενική Διεύθυνση ε, για τη Δικαιοσύνη, DG Justice, ε, θεωρήθηκε ότι ήταν κυρίως θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν καταλαβαίνω γιατί μεταφέρθηκε τώρα από την Γενική Διεύθυνση Justice στην Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση. Αλλά έτσι νομίζω ότι χάνουμε πολλές ευκαιρίες με τη μεταφορά αυτή, διότι δεν μπορούμε να ε, ε, έχουμε την διατομιακή οπτική στα δικαιώματα, διότι στην Γενική Διεύθυνση Justice έχουμε τα δικαιώματα ε, ηλικιωμένων, γυναικών, διεμφυλικών κλπ. Όχι όμως των ατόμων με αναπηρία. Αυτά τα δικαιώματα έχουν μεταφερθεί στη Γενική Διεύθυνση για την Επασχόληση και νομίζω ότι αυτό στέλνει αρκετά αρνητικό μήνυμα Ωστόσο υπάρχει και μια θετική πλευρά. Νέος αντιπρόεδρος σας ε, θα μπορούσε να είναι το νέο σημείο εστίασης ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα στείλει ακόμα πιο ισχυρό μήνυμα όσον αφορά την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, υπάρχουν ε, τρεις ε, φορείς, το κράτος, ο ανεξάρτητος μηχανισμός παρακολούθησης και η φωνή των ανθρώπων με αναπηρίες. Τη συμμετοχή αυτή την επικροτούμε με κάθε τρόπο, είτε έχει να κάνει με το συντονισμό, με τα σημεία με τη συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους Αλλιώς ε, δεν θα υπάρξει πλήρης εφαρμογή της ε, σύμβασης. Θα ήθελα λοιπόν ε, να φροντίσουμε να ακούγεται η φωνή των ανθρώπων με αναπηρίες και κατά την εφαρμογή και κατά την παρακολούθηση και εντός του δικτύου σας για τη σύμβαση και επίσης να υπάρχουν επαρκείς πόροι. Και η τελική μου παρατήρηση αφορά το άρθρο 32. Όπως ανέφερα, ε, είναι αρκετά ισχυρή η διατύπωση στις συστάσεις μας σχετικά με το άρθρο 32. Λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ε, ανθρωπιστικής βοήθειας σε διεθνές επίπεδο. Έτσι λοιπόν έχει μοναδική θέση και μπορεί έτσι να κατέχει ηγετική θέση στην εφαρμογή των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω στις εξωτερικές σας δράσεις να φροντίσετε να έχετε αναλυμένα δεδομένα και να δείξετε στον κόσμο τι αλλαγές μπορούμε να επιφέρουμε συμπεριλαμβάνοντας τα δικαιώματα ανθρώπων με αναπηρίες σε όλες τις ε, εξωτερικές δράσεις. Ε, θα κλείσω εδώ. Θα είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω μέσω στο λόγο στον κύριο Μάικλο Φλάχερτη, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ο οποίος είναι διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Παρακαλώ. Thank you, Mr. Madam Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Εισηγήτρια, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί φίλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε σήμερα να συμμετάσχω σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για το ζήτημα αυτό σήμερα το πρωί. Ζήτημα πολύ σημαντικό έχουμε πολύ σημαντικές προτεραιότητες. Πρώτον, πλησιάζει η δέκατη επέτειος της σημαντικότητας αυτής σύμβασης των ΗΠΑ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Προχωράμε αυτή τη στιγμή σε μία, από μία ιατρική προσέγγιση των ατόμων με αναπηρία σε μία προσέγγιση που εστιάζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην κατάργηση οποιασδήποτε διάκρισης κατά των ατόμων αυτών. Δεύτερον, εξίσου σημαντικό, είναι ότι έχουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσχωρήσει στη σύμβαση αυτή. Πρώτη φορά στην ιστορία της σύμβασης αυτής έχουμε μια περιφερειακή οργάνωση η οποία προσχωρεί στη σύμβαση αυτή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η εφαρμογή μπορεί να γίνει πολύ καλύτερα κατά αυτόν τον τρόπο. Τρίτο σημαντικό, για πρώτη φορά έχουμε μια σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών η οποία ουσιαστικά μπορεί να, κάνει, να προχωρήσει σε συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων λοιπόν αυτών και κατά αυτόν τον τρόπο μας δίνεται μια πολύ σημαντική ευκαιρία να τα αντιμετωπίσουμε σωστά. Τέταρτον, απευθύνομαι σήμερα στην Επιτροπή σας στα πλαίσια του πλαισίου παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 33 της Σύμβασης και βλέπετε ότι εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συμμετέχουν. Έχουμε το κοινοβούλιο το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ο Ευρωπαίος και Μεσολαβητής, ο οποίος ελέγχει το πώς εφαρμόζεται η σύμβαση αυτή, τον Οργανισμό Θεμελιδών Δικαιωμάτων, καθώς επίσης και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ατόμων με Αναπηρία που συμμετέχει και αυτό ισότιμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι καταφέρνουμε να εμπλέξουμε όλους αυτούς τους φορείς στο πλαίσιο παρακολούθησης ε, της σύμβασης ε, CRPD όπως μας, την, ε, μας το περιέγραψε η κυρία Στίβενς. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης κύριε Πρόεδρε το ότι διεξάγεται μία ακρόαση όσον αφορά τα καταληκτικά συμπεράσματα της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων Αναπηρία. Για άλλη μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματικά θέτει ένα πολύ θετικό παράδειγμα. Όσον αφορά τις συγκεκριμένε αυτές ε, καταληκτικές συστάσεις, ξέρετε ότι πρόσφατα καταλήξαμε σε αυτές στα πλαίσια της Επιτροπής CRPD. Μιλάω όπως βλέπετε στα αγγλικά, και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω ένα όρο. Από το Keeper περνάμε στο poacher. Δηλαδή, εγώ για 8 χρόνια συμμετείχα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπου μπορούσαμε και εκεί να καταλήξουμε σε κάποιες συστάσεις και συμπεράσματα που απευθύνονταν προς τα κράτη-μέλη. Μπορώ λοιπόν να πω ότι πραγματικά έχω συσσωρεύσει μια πολύ θετική εμπειρία από την δραστηριότητα αυτή έχοντας ένα διαφορετικό ρόλο στο παρελθόν. Αν δείτε λοιπόν τις καταληκτικές παρατηρήσεις και το σχετικό αυτό έγγραφο, έχουμε 94 τέτοιες συστάσεις. Το έγγραφο αυτό φαίνεται αρκετά φορτικό, αρκετά βαρύ θα έλεγα, αλλά αν εξετάσουμε τις συστάσεις αυτές μία προς μία, θα δείτε ότι είναι πραγματικά πολύ σωστά διατυπωμένες, αντλούν πληροφορίες σε πολλές διαφορετικές πηγές και θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα εύστοχες. Πραγματικά φαίνεται στις συστάσεις αυτές ποιο είναι το πρόβλημα και πώς μπορεί να λυθεί μέσω συγκεκριμένων πολιτικών συστάσεων, μέσω συγκεκριμένης ανάληψης δράσης. Τούτων λεχθέντων βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι δεσμευτικές αυτές οι συστάσεις. Οι συστάσεις αυτές δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση κάποια δεσμευτική οδηγία προς τα κράτη-μέλη. Ουσιαστικά απευθυνόμαστε προς τα κράτη-μέλη και προκειμένου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Επίσης, οι συστάσεις αυτές δεν είναι απολύτως δεν είναι τέλειες. Ξέρετε ότι ε, ένα όργανο παρακολούθηση ε, των ε, Ηνωμένων Εθνών δεν μπορεί να γνωρίζει απόλυτα ποιε είναι οι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ακριβώ, διαβάζοντα τι συστάσει αυτέ, ποιε απευθύνονται περισσότερο στα κράτη-μέλη και ποιε συστάσει απευθύνονται περισσότερο στην κοινοτική αρμοδιότητα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα θα μπορούσαν να διατυπωθούν και καλύτερα οι συστάσει αυτέ. Για παράδειγμα, η σύσταση 50 που είχε να κάνει με το άρθρο 43 ουσιαστικά προκαλεί μια σύγχυση ανάμεσα στο ρόλο της παρακολούθησης και στο ρόλο της εφαρμογής. Και νομίζω ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν εδώ πέρα οι αρχές των Παρισίων, πέρα από τα όσα λέγονται δηλαδή για το άρθρο 33. Νομίζω ότι αν αφήσουμε πάντως εκτός αυτά τα μικροπροβλήματα, έχουμε ένα πολύ κατάλογο συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον οποίο πρέπει να λάβουμε απόλυτη σοβαρότητα. Πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, θα ήθελα λοιπόν να επικεντρωθώ σε τρει συγκεκριμένε συστάσει στην παρουσίασή μου αυτή. Πρώτον, θα ήθελα να φερθώ στην παράγραφο 11 των παρατηρήσεων αυτών, όπου λέμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία για την περίοδο 2010 με 2020. Μας δίνεται λοιπόν εδώ η ευκαιρία να κάνουμε έναν απολογισμό να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι δεσμεύσεις που αναλάβαμε το 2010, να καταφέρουμε να δούμε ποιες είναι οι σχετικές συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών και να καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να εντοπίσουμε νέους δείκτες και να καταφέρουμε να εστιαστούμε περισσότερο στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα ήθελα συνέχεια να περάσω στην παράγραφο 50 όπου έχουμε μια πολύ σημαντική διάταξη που αναφέρεται στην αυτόνομη ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία. Λέγεται εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προχωρήσει σε δράσεις από ιδρυματοποίησης και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθούν τα ευρωπαϊκά διατροτικά και επενδυτικά ταμεία προκειμένου να προωθηθούν αυτές οι δράσεις από ιδρυματοποίησης. Νομίζω ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και ελοχεύουν εδώ πέρα κάποιοι κίνδυνοι να καταφέρουμε τελικά να αποκριθούμε στι ε, προκλήσει που τίθενται ενώπιον μα. Ο δικό μου οργανισμό, ο Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να βοηθήσει τι δράσει αυτέ αποδρυματοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από τον επόμενο μήνα, όπου θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα από την επιτόπου εργασία που έχουμε κάνει σε διάφορα ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε πώς οι άνθρωποι που βγαίνουν από τα ιδρύματα αυτά μπορούν να ενταχθούν στη συνέχεια στην ε, κοινωνία. Τέλος, όσον αφορά τις ε, συστάσει που έχουν να κάνουν με το πλαίσιο παρακολούθησης σύμβασης, να επαναλάβω κάποια σημεία τα οποία έθιξε η κυρία Στίβεν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το πλαίσιο αυτό παρακολούθησης να ενισχυθεί όχι μόνο μέσω της εγγύηση ανεξαρτησία του, αλλά να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε και ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο το οποίο να έχει και τους απαραίτητους πόρους, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή όλα τα μέλη, το κάθε μέλος ξεχωριστά του πλαισίου αυτού, εναπόκειται στους δικούς του πόρους, προκειμένου να καταφέρει να συμμετέχει αποδοτικά στο πλαίσιο αυτό παρακολούθησης. Ολοκληρώνοντας λοιπόν κύριε Πρόεδρε, ας θυμηθούμε ότι οι συστάσεις αυτές, οι καταληκτικές, αποτελούν μέρος μιας κυκλικής διαδικασίας η οποία συνεχίζεται παόριστον. Έχουμε λοιπόν αυτές τις καταλεκτικές συστάσεις, περνάμε πλέον στη φάση της εφαρμογής. Η φάση λοιπόν αυτή της εφαρμογής θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια συνεχούς διαλόγου με τους βασικούς ενδιαφερομένους φορείς, ιδίως με τα άτομα τα οποία ζουν με αναπηρίες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια συνεχής δέσμευση των ανθρώπων αυτών με το πλαίσιο παρακολούθησης. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο, μόνο μέσω της συνεργασίας αυτής θα καταφέρουμε σε μερικά χρόνια να υποβάλουμε μια νέα έκθεση στην Επιτροπή των ΕΕ και θα καταφέρουμε να λάβουμε από την Επιτροπή αυτή τα νέα καταληκτικά συμπεράσματα. Προφανώς εκείνη τη χρονική στιγμή δεν θα έχουμε υλοποιήσει και τι 94 συστάσεις. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το πιο σημαντικό είναι να καταφέρουμε καλή την πίστη, να δεσμευτούμε για την εφαρμογή ορισμένων από τις συστάσεις αυτές, έτσι ώστε την επόμενη φορά, στην επόμενη έκθεση, οι νέες συστάσεις που θα μας δώσει η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση εφαρμογής. Εξ αρχής είχα πει, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουμε πέντε σημαντικές, σημαντικότερες πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη CRPD. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι θα καταφέρουμε πέρα από τις σημαντικές αυτές της πρωτοβουλίες να προχωρήσουμε και στη θέσπιση καλών πρακτικών συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να προωθήσουμε τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία παντού στην Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ενδιάμεση παρατήρηση. Αυτή η κίτρινη κάρτα που έβγαλα δεν ήταν τεστ. Ε, ήταν μια παρέμβαση Ε, στο Αμβούργο υπάρχει μια κυρία η οποία πρέπει ε, όλα αυτά να τα μεταφράζει σε αυτό που βλέπετε ε, εδώ σε αυτή την οθόνη. Και επειδή μιλούσατε πάρα πολύ γρήγορα, σας έβγαλα την κίτρινη κάρτα. Γιατί είναι δύσκολο κανείς να μεταφράζει και να τα γράφει για να τα βλέπετε εσείς ε, στην οθόνη. Λοιπόν, το λόγο έχει κύριο ο Ράιλι, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κυρίες και κύριοι. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Σέβενς, Ευρωβουλευτή, που με κάλεσε να συζητήσουμε την εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ και ιδιαίτερα τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία. Ως εποπτικό όργανο, ο διαμεσολαβητής έχει ιδιαίτερη ευαισθησία για την ανάγκη να ακούμε τι έχει να μας πει ο ΟΗΕ και η Επιτροπή για το πώς συμμορφούνται ή δεν συμμορφούνται η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη σύμβαση αυτή. Συχνά έχω πει ότι τα δικαιώματα καλύπτονται από συμβάσεις, χάρτες και σε θεσμικό πλαίσιο και μάλιστα αυτά τα έχουν και στους ε, κορνιζωμένα, αλλά αυτά είναι οδικοί χάρτες, δεν είναι διακόσμηση για τους τείχους των θεσμικών οργάνων. Πολλά παραμένουν ευκολόγια, αλλά τα ευκολόγια αυτά είναι κάτι που αφορά την καθημερινή ζωή ατόμων με αναπηρία και τα μετράνε και τα βλέπουν στη ζωή τους η κυρία Κίξτον και άλλοι συνάδελφοι της Επιτροπής του ΟΗΕ έχουν αξιολογήσει τους κανόνες, τις ε, συμπεριφορές και ε, τις συνήθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δικό μου γραφείο έχει αρχίσει να υλοποιεί τις παρατηρήσεις ε, της Επιτροπής αυτής. Σύμφωνα με τη σύμβαση λοιπόν, βασική μου υποχρέωση είναι να προστατεύω τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να διεκπεραιώνω τις καταγγελίες και τα παράπονα που φτάνουν στα χέρια μας και αφορούν τα θεσμικά όργανα, του οργανισμού, τους φορείς της Ένωσης. Οποιοδήποτε πολίτης ή άλλος άνθρωπος που διαμένει στην Ένωση, φυσικό πρόσωπο είτε και νομικό πρόσωπο που έχει έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποβάλει καταγγελία. Ο καταγγέλων δεν χρειάζεται προσωπικά να έχει φυγεί από την ε, ε, εικαζόμενη κακοδιαχείριση ή να έχει νομική ε, αρρωγή δικηγόρο να τον εκπροσωπεί. Ορισμένε καταγγελίες αφορούν την πρόσβαση των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, των κτηρίων δηλαδή. Ένας υπάλληλο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αναπηρικό αμαξίδιο ε, ισχυρίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν του παρέχει επαρκή πρόσβαση στο χώρο εργασία του. Άλλο λέγει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν κάνουν ό,τι πρέπει ε, ως διαβήματα στις τοπικές αρχές για να υπάρχουν αρκετές θέσεις αναπήρων ε, για στάθμευση κοντά ε, στα κτίρια. Καμιά φορά δεν υπάρχει διερμηνία στην νοηματική γλώσσα σε βασικά θέματα και σε διοργανώσεις. Σε κάποια περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάστηκε να αποζημιώσει ε, κάποιον ενδιαφερόμενο ή να δεσμευτεί ότι θα έχει νοηματική γλώσσα σε μελλοντικέ διοργανώσει. Ε, άλλοι πολίτε ε, λέγουν ότι έχουν δυσκολίε να επικοινωνούν με τα θεσμικά όργανα γιατί δεν έχουν την απαραίτητη πληροφόρηση σε τρόπο τον οποίο μπορούν να τη διαβάσουν. Ένα καταγγέλων είπε ότι ο διαδικτυακός τόπος Europass για να υποβάλει κανείς το βιογραφικό του στο διαδίκτυο δεν έχει πρόσβαση για άτομα με αναπηρία και μάλιστα ε, για τους τυφλούς. Στο γραφείο μου προσεχώς έχουμε κατάρτιση ε, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι τα έντυπα και τα ενημερωτικά φυλάδια που στέλνουμε στους ενδιαφερομένους ε, είναι σε θέση ήδη να τα διαβάζουν. η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι υποδειγματική και να αυξάνει την απασχόληση ατόμων με αναπηρία σε όλα τα θεσμικά όργανα. Και υπήρξε μια περίπτωση ενό ατόμου που είχε πρόβλημα στην ακοή και έκανε μια καταγγελία. Ε, ε, παρόλο που έχει καλό μητρό και καλέ επιδόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι καταγγελίε που λαμβάνουμε και έχουν να κάνουν με αναπηρίε δυστυχώ ε, είναι περιορισμένε αυτό το καιρό ψάχνουμε πώς μπορούμε να προβάλλουμε καλύτερα τον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή έτσι ώστε να μπορούν να αποτείνονται σε εμά άνθρωποι που μας χρειάζονται γιατί δεν μας γνωρίζουν. Ξέρω ότι πολλοί από εσά είστε μόνοι με επαφή με ψηφοφόρους σας από την εκλογική σας περιφέρεια που μπορεί να μας χρειάζονται και παρακαλούμε βοηθήστε μας να διαδοθεί η είδηση ότι υπάρχει ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής. Από τότε που ανέβαλα ε, όπως θα γνωρίζετε, έχω κάνει στρατηγικές μελέτες για να αντιμετωπίσουμε συστημικά προβλήματα και ελλείψεις στα θεσμικά όργανα. Μία έρευνα κοίταξε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πολιτική Συνοχή έτσι ώστε να συνάδει με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, τα χρήματα χρησιμοποιούνται για να ε, μπαίνουν σε ιδρύματα οι άνθρωποι με αναπηρία αντί να τους βοηθούμε να εντάσσονται στην κοινωνία έκλεισα με 8 κατευθυντήρες γραμμές και προτάσεις στην έρευνα αυτή ε, για ε, να επιβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη-μέλη και να κάνει ελέγχους επιτόπου με επισκέψεις στα κράτη για να ε, δουν πώς εφαρμόζουν τα προγράμματα συνοχής. Θα πρέπει επίσης να λασάρει μια πλατφόρμα online όπου μπορεί η κοινωνία των ε, πολιτών να καταγγέλει παραβιάσεις του χάρτη του ΟΗΕ για ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα στη χρήση των κονδυλίων. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι αυστηρότατη και να πεί πτυράβδος όταν τα κράτη-μέλη δεν τηρούν τις υποχρεώσεις του. Θα πρέπει να ελέγχει ότι λειτουργούν σωστά οι μηχανισμοί ανάκτησης κονδυλίων και αποζημίωσης στα κράτη-μέλη και να φροντίζει να μην γίνονται αυτές οι παραβιάσεις με κατάρτιση, με εκπαίδευση, με δυνατότητες στα κράτη-μέλη που υστερούν ε, στη συγκεκριμένη υπόθεση. Χάρηκα που έδωσε συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έρευνα. Την έρευνά μου αυτή θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Πρόσφατα ε, ιδρύθηκε μια μονάδα για στρατηγικές ε, μελέτες και έρευνες στο γραφείο μας, έτσι ώστε στο μέλλον να ασχολείται με ειδικά θέματα. Και βεβαίως... Ε, Εκεί έχουμε και τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ. Αυτό που μας ε, προβληματίζει αυτό το καιρό είναι η πρόσβαση στις ισοσελίδες των θεσμικών οργάνων. Η Επιτροπή του ΟΗΕ έχει εντοπίσει προβλήματα και ελλείψεις που πρέπει να διορθώσουμε. Έστειλα μια επιστολή πρόσφατα στον πρόεδρο Γιούνκερ, καθώς τα περισσότερα όργανα, ε, οργανισμοί ε, και λοιποί φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στρέφονται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, πάρουν το παράδειγμα. Θα πρέπει η ιστοσελίδα τους να είναι πιο φιλική προς το χρήση και πιο προσβάσιμη. Με την υποστήριξη ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων έχουμε στην ιστοσελίδα μας 24 γλώσσες σχετικές οδηγίες. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Το κείμενο έχει και εικόνες και θα το δημοσιεύσουμε ε, προσεχώς και εμείς ήδη έχουμε περισσότερα να κάνουμε. Η δική μου εντολή δεν μου επιτρέπει να εργαστώ ε, επί όλων των καταληκτικών παρατηρήσεων. Ας πούμε, τα ευρωπαϊκά σχολεία είναι εκτός της δική μου εντολής. Αλλά επειδή ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα και τα έχει εντοπίσει η Επιτροπή, προσπάθησα εγώ να έρθω σε ένα επικοδομητικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων και τα χρηματοδοτεί κιόλας εν μέρη Έστειλα και μια επιστολή στην Αντιπρόεδρο Γεωργίευα τον περασμένο μήνα. Επίση, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μα η επιστολή αυτή. Οι καταληκτικέ παρατηρήσει, λοιπόν, ω προ το πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ ανησυχητικέ. Όχι απλώ επειδή εντοπίζουν κάποια προβλήματα και κάποιε προτεραιότητε, αλλά όποιο και να είναι το πλαίσιο, πάντα θα πρέπει να εντάσσεται και να υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής των Μένων Εθνών. Γι' αυτό χρειάζεται τεχνική βοήθεια, η παροχή τεχνικών συμβουλών ε, από την Επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα από ό,τι κατάλαβα στα πλαίσια της σύμβασης. Στο μεταξύ σας παρακαλώ να βεβαιωθείτε ότι το γραφείο μου θα συνεχίσει να αυξάνει τη συνειδητοποίηση για τη δυνατότητα ε, υποβολής καταγγελιών και παραπώνων που έχουν να κάνουν με άτομα με αναπηρία και καταχρήσεις θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα στρεβλά στο μέλλον, γιατί είμαστε προσιλωμένοι και αποφασισμένοι στην υπόθεση αυτή. Να προστατεύσουμε κάθε πολίτη της Ένωσης, κάθε άτομο με αναπηρία που θα πρέπει να έχει γνώση των δικαιωμάτων και των ε, δυνατοτήτων του. Ευχαριστώ πολύ. Κατόπιν ε, έχουμε την ε, Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ ε, των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, κυρία Γκούντα Άγκα. Καλημέρα σε όλους. Θα μιλήσω λετονικά. Mm. Παρακαλώ λοιπόν φορέστε τα ακουστικά σας. Βρίσκομαι σήμερα εδώ και εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και χαίρομαι πολύ που μπορώ να εκπροσωπώ αυτόν τον μεγάλο οργανισμό που καλύπτει μια σειρά οργανισμών ε, εθνικών και ευρωπαϊκών. Έχουμε επίσης εταίρους και είμαι βέβαιη ότι οι πολλές διαφορετικές οργανώσεις ε, που βρίσκονται υπό την αιγύδα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μας επιτρέπει να παρουσιάσουμε έγκυρα τις απόψεις ε, των ε, ανθρώπων με αναπηρία. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να ανταλλάξουμε απόψεις με τους ευρωβουλευτές. Οι συστάσεις που αναφέρθηκαν στις ομιλίες των προλαλισάντων είναι ιδιαίτερα σημαντικές ε, και για μας, ε, για το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι η εξής. Κυρία Στίβενς, σας ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που έχετε κάνει. Η παρουσία μας εδώ σήμερα για να συζητήσουμε το θέμα αυτό μας δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει σωστά το άρθρο 4.3 που λέει ότι είναι πολύ σημαντική η γνώμη των ε, οργανώσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες και θα πρέπει να συμμετέχουν οι οργανισμοί αυτοί στην ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα διότι θέλουμε να παρουσιάσουμε τη θέση μας ε, στη συζήτηση αυτή. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ ε, Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες εκτιμάει το δίκτυο που έχει δημιουργήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της σύμβασης ε, του ΟΗΕ. Πιστεύουμε ότι είναι ζωτικό αυτό για να εφαρμοστεί πλήρως η σύμβαση. Δυστυχώ, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ατόμων με ειδικέ ανάγκε δεν συμμετέχει άμεσα στο δίκτυο αυτό. Αλλά μάλλον ως διαμεσολαβητής και ως μέρος του δικτύου παρακολούθησης. Ωστόσο πιστεύουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Σύμβασης ε, θα ήταν σημαντικό το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες να ε, συμμετέχει άμεσα στο δίκτυο αυτό. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ε, θεωρεί ότι Χρειάζεται πιο δομημένος διάλογος ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους ανθρώπους με αναπηρίες. Η Επιτροπή του ΟΗΕ αναφέρει ακριβώς αυτόν τον διάλογο και για να βελτιωθεί ο διάλογος αυτός, να δομηθεί περισσότερο, η οργάνωσή μας εκπονεί συστάσεις σχετικά με τη μορφή που θα μπορούσε να έχει αυτός ο διάλογος. Ε, και επίσης ε, σχετικά με το πώς ε, μπορεί να οργανωθεί καλύτερα αυτός ο διάλογος. Θα ήθελα εδώ να τονίσω κάποια σημαντικά στοιχεία. Καταρχάς, Θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντική είναι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι μπορεί να δείξει ότι ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ηγηθεί στην ε, διαδικασία εφαρμογής των συστάσεων της Επιτροπής του ΟΗΕ. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος περιφερειακός οργανισμός χωρών που εφαρμόζει μια τέτοια σύμβαση. Είναι η πρώτη περιφερειακή δομή που έχει λάβει τέτοιες συστάσεις και αυτό Ε, σημαίνει ότι έχετε και μεγάλη ευθύνη σχετικά με την ε, εφαρμογή των συστάσεων και θα ήθελα να αναφέρω διάφορες πτυχές. Καταρχάς, ε, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτομα με αναπηρίες για το διάστημα 2010 με 2020. Συζητάμε εάν έχει εφαρμοστεί σωστά η στρατηγική αυτή. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ θεωρεί ότι η κατάρτιση της ε, στρατηγικής στο μέλλον, ε, καθώς και η διατύπωση συστάσεων εντός της στρατηγικής ε, μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο, διότι πρέπει να εφαρμοστούν οι συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ. Η στρατηγική αυτή μπορεί να βελτιωθεί μόνο σε στενή συνεργασία με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι απόψεις των ανθρώπων αυτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασχοληθεί με την αξιολόγηση της πολιτικής και να δει τα πάντα μέσα από το πρίσμα αυτής της σύμβασης για να εξετάσει αν έχουν ληφθεί υπόψη οι συστάσεις. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για την ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα που βασίζεται ε, στην αρχή της ε, ενιαίας αγοράς. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική νέα πρόταση ε, στην ιστορία της Ευρώπης. Καταρχάς μιλάμε για προσβασιμότητα ανθρώπων με αναπηρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά στο άρθρο 9 της σύμβασης ε, βλέπουμε ότι η πράξη αυτή δεν αναφέρεται στο άρθρο 9. Δυστυχώς ε, το θέμα της ε, προσβασιμότητας δεν εξετάζεται. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις. Υπάρχουν και πολλές άλλες νομικές πράξεις τις οποίες θα πρέπει να επανεξετάσουμε. Θέλουμε οι ιστοσελίδες ε, να είναι πιο εύκολα προσβάσιμες ε, και Η διαμεσολαβήτρια ανέφερε ότι κάποιες ε, ιστοσελίδες είναι μόνο εν μέρη ή καθόλου προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρίες. Επίσης, οι αναπηρίες δεν επιτρέπεται να αποτελούν λόγο διάκρισης. Άλλωστε έχουμε την ε, σύμβαση Μαρακές Κωνσταντινούπολης ε, και Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα έχουμε βοήθεια για την εφαρμογή ε, των νομικών αυτών πράξεων. Θα ήθελα επίσης να τονίσω μια άλλη σημαντική σύσταση της Επιτροπής του ΟΗΕ. Αναφέρομαι στην ελάχιστη κοινωνική προστασία ανθρώπων με αναπηρίες. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η κρίση και τα μέτρα λιτότητας, οι μεγάλες περικοπές στον προϋπολογισμό, έχουν επιδεινώσει την κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες σε πολλές χώρες. Πολλές χώρες ε, θεωρούν ότι τα σχετικά μέτρα είναι πολύ δαπανηρά. Γι' αυτό προτιμούν ε, να τοποθετούνται τα άτομα με αναπηρίες σε ιδρύματα, θεωρούν ότι είναι πιο οικονομική επιλογή. Αλλά έτσι χάνουμε την ευρύτερη εικόνα. Το πώς δηλαδή όλα αυτά επηρεάζουν ε, την καθημερινή ζωή ανθρώπων και το θέμα της κοινωνικής προστασίας. Είμαστε ευγνώμονες που τα Διαστατικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες σε υπηρεσίες. Καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φροντίσει όλα να εξετάζονται υπό το πρίσμα της σύμβασης του ΟΗΕ. Κατά τη γνώμη μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής του ΟΗΕ. Φαίνεται φιλόδοξο σχέδιο αυτό. Το να λέμε ότι όλοι είναι ίσοι εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, άσχετα με το ε, εάν κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποιε αναπηρίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τώρα τον ε, εκπρόσωπο του ΟΗΕ, τον κύριο Γιάννη. Παρακαλώ. Ladies and gentlemen, I would like... Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, πρόσκληση που απίφθινε στην ύπατη αρμοστία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τον κεντρικό ρόλο που έχει αναλάβει για το ζήτημα αυτό. Να ξεκινήσω καταρχά λέγοντα κάποια πράγματα όσον αφορά τον ρόλο που διδραματίζει η ύπατη αρμοστία ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδίω σε σχέση με την ε, Επιτροπή των ΗΕ για τα Δικαιώματα των με Αναπηρία που βέβαια λειτουργεί αυτόνομα. Εμείς ε, στην Γενέβη παρέχουμε διοικητική υποστήριξη προς διάφορες επιτροπές των Ηνωμένων και προς συγκεκριμένη αυτή επιτροπή και βέβαια υποστηρίζουμε και το έργο του ε, εισηγητή για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και έχουμε και ένα γραφείο εδώ στις Βρυξέλλες που καλύπτει την συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εργαζόμαστε εδώ πέρα για την εκπροσώπηση της Επιτροπής αυτής, για την προώθηση το έργο των διαφόρων επιτροπών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και προωθούμε προφανώς και την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής CRPD των Ηνωμένων Εθνών και συνεργαζόμαστε επίσης και με την κοινωνία των πολιτών καθώς επίσης και με εθνικά, εθνικούς φορείς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνεργαζόμαστε επίσης με τις αρμόδιες αρχές τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφορά δηλαδή τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκής Ένωση, προσπαθούμε να συμβάλλουμε και εμείς στο σχεδιασμό κοινοτική πολιτική, αλλά και με τα επιμέρου κρατη κράτη-μέλη και μαζί με το EDF, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, συμμετέχουμε σε μια ομάδα πυρογνωμόνων για την μετάβαση από τα ιδρύματα προς την κοινωνία, για τις δράσεις δηλαδή από ιδρυματοποίησης. Αναφέρθηκαν ήδη από τις προελίσσαντες ορισμένες σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και όλες αυτές οι προκλήσεις εμφανίζονται στις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών. Να αναφερθώ σε κάποιες από αυτές μόνο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά άτομα αναπηρία που βρίσκονται σε ιδρύματα σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετική αναφορά γίνεται σε πάρα πολλές συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών. Το θέμα δεν έχει να κάνει μόνο με το άρθρο 19, δηλαδή με την αυτόνομα ανεξάρτητη διαβίωση των ανθρώπων αυτών, αλλά έχει να κάνει και με ένα πολύ θεμελιώδες δικαίωμα των ανθρώπων αυτών προκειμένου να μπορούν να χαίρουν και άλλων δικαιωμάτων τους. Και πολύ συχνά βλέπουμε το ζήτημα αυτό να συνδυάζεται με την έλλειψη κάποιας νομικής ικανότητας. Άρθρο 12 όσον αφορά δηλαδή την δικαιοπρακτική ικανότητα των ατόμων αυτών. Βλέπουμε ότι η κατάσταση διαφέρει από τη μία χώρα στην άλλη όσον αφορά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για την έξοδο από τα ιδρύματα και την πιο αυτόνομη ζωή. Επίσης, δεν υπάρχει απαραίτητη πρόσβαση σε ορισμένες ε, συμβατικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτή αγορά εργασίας πάλι χωρίς διακρίσεις και χωρίς αποκλεισμούς και γενικά πρόσβαση σε διάφορες πτυχές εκφάνσεις της ε, ζωής και της συμμετοχής στα κοινά. Και βέβαια έχουμε και τις επιπτώσεις των πολιτών λιτότητος στη ζωή των ανθρώπων με αναπηρίες. Αυτό ήδη αναφέρθηκε από κάποιον προαλήσαντα. Η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε πραγματικά να συμβάλλει στην ε, καλύτερη διαβίωση των ανθρώπων με αναπηρία στα κράτη-μέλη της Ένωσης και εμείς θα θέλαμε να πούμε ότι ε, μπορεί να το κάνει αυτό πέρα από τους τομείς αρμοδιότητάς της. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εγκρίνει σχετική νομοθεσία ή να ολοκληρώσει νομοθεσία που αυτή τη στιγμή εκκρεμεί, όπως για παράδειγμα η νέα πράξη προσβασιμότητας ή η παλαιότερη πρόταση όσον αφορά την οριζόντια αυτή οδηγία για την κατάργηση των διακρίσεων ζητήματα τα οποία αναφέρονται και τα δύο σκαταληκτικέ παρατηρήσει τη Επιτροπή, αλλά θα μπορούσε επίση η Ευρωπαϊκή Ένωση να ερμηνεύσει την νομοθεσία κατά τρόπον τέτοιο ώστε οι υφιστάμενες κοινοτικέ νομοθεσίες, οι υφιστάμενοι κοινοτικοί νόμοι να εφαρμόζονται σωστά από τα κράτη-μέλη, να συνάδουν δηλαδή με τις αρχές της σύμβασης αυτής και θα μπορούσε βέβαια να προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα, είτε αυτά τα οποία θα μπορούσαν να έρθουν κατευθείαν από τις Βρυξέλλες, είτε αυτά που συγχρηματοδοτούνται με τα κράτη-μέλη. Βλέπετε εδώ πέρα στην εικόνα τον ε, καθηγητή Jerome Quinn, ένας από τους βασικούς ιδρυτές της σύμβασης, ο οποίος εδώ πέρα βλέπετε ότι να φέρει κάτι το οποίο εμφανίζεται σε μια δημοσίευση της δικής μας, του δικού μας του γραφείου και στη φράση αυτή βλέπετε ότι η κοινή αυτή μεταχείριση και διαχείριση δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει κάποια ευθύνη για τη διαχείριση των πόρων αυτών των χρηματοδοτικών μέσων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί σίγουρα έχει σημειωθεί πολύ σημαντική πρόοδος από τη μία πλευρά. Βλέπουμε ότι η χρηματοδότηση, τα απαραίτητα αυτά κονδύλια έχουν βοηθήσει όντως τις δράσεις της αποδρυματοποίησης σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα όμως βλέπουμε ότι μολονότι έχουμε κάποιες θετικές αλλαγές και θετικές προσαρμογές, γίνονται από την άλλη επενδύσεις οι οποίες είναι ουσιαστικά επιφανειακές ενώ δεν αλλάζει τελικά το ίδιο το μοντέλο το οποίο θα πρέπει να ακολουθούμε. Βλέπετε εδώ πέρα μια εικόνα από την δική μου τη χώρα, την Τσεχία, μια φωτογραφία η οποία, την οποία βγάλαμε πριν από 7 περίπου χρόνια, όταν αρχίσαμε να ενδιαφερόμαστε περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δράση της ε, σύμβασης αυτής και ουσιαστικά εδώ πέρα αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε είναι ότι θέλουμε να αλλάξουμε το μοντέλο αυτό το οποίο βλέπετε να απεικονίζεται με τη φωτογραφία αυτή στην ε, διαφάνεια την οποία σας δείχνω. Ακριβώς τη δράση λοιπόν αυτή, την ενεργή θέλουμε να αναλάβουμε και πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο καλείται να επιβλέπει τη δράση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με δράσεις ιδρυματοποίησης ή και άλλες δράσεις. Οι πόροι αυτοί λοιπόν θα πρέπει να προωθούν την δυνατότητα των ανθρώπων αυτών να ζουν μέσα στην κοινωνία, να μην περνάνε απλώς από μεγάλα ιδρύματα σε μικρότερα ιδρύματα, να μην διονύζεται δηλαδή αυτό το μοντέλο της Επίσης, επίσης, θέλουμε και δράση στον τομέα της απασχόλησης. Πέρα από τα όσα λέει ρητά η σύμβαση, νομίζω ότι ήδη η ε, Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών αλλά και η απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει αυτή τη στιγμή μας δείχνει τι μπορεί να λειτουργήσει και τι όχι ως δράση για την καλύτερη ένταξη των ανθρώπων αυτών στην αγορά εργασίας. Και βέβαια θα πρέπει να προωθήσουμε εδώ πέρα τα θετικά παραδείγματα, τις θετικές δράσεις, αυτές που έχουν οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε τις δράσεις ε, απασχόλησης δηλαδή να συνεργαστούμε με τους εργοδότες και να καταφέρνουμε να προωθούμε την πρόσληψη των ατόμων με αναπηρίες σε ποιοτικέ δουλειές, με σωστές αποδοχές, σωστή δηλαδή και ολοκληρωτική ένταξη στην αγορά εργασίας και να μην προωθούμε απλώς την πολύ περιορισμένη εργασία τους σε κάποια εργαστήρια χωρίς τα άτομα αυτά να έχουν κάποια προοπτική στη συνέχεια να αποκατασταθούν σε μια θέση απασχόληση, σε μια μόνιμη θέση απασχόληση. Δεν θέλουμε απλώ τα άτομα αυτά να λαμβάνουν κάποια πιστοποιητικά ότι έχουν απασχοληθεί σε κάποια εργαστήρια. Θέλουμε επίση να μπορούν να συμμετέχουν τα άτομα αυτά περισσότερο σε προγράμματα κατάρτιση και εκπαίδευση. Α περάσουμε τώρα λίγο πέρα από την νομοθεσία και πέρα από τα χρηματοδοτικά μέσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λάβει δράση και σε άλλου τομεί. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στου τομεί εκείνου όπου μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να νομοθετήσει ίσως τομεί εκείνους που μπορεί να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον έναν άλλο τρόπο. Υπάρχουν και άλλοι τομείς στου οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωση μπορούν να αναλάβουν δράση. Για παράδειγμα, και στον τομέα αυτό, στον τομέα του συντονισμού και της πολιτικής ηγεσία. Ξέρετε ότι υπάρχει μια στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία, Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα αναθεωρηθεί η στρατηγική αυτή γιατί μπορεί να γίνει πιο φιλόδοξη. Η είπατε αρμοστία των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα λυπάται αυτή τη στιγμή που η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως διαμορφώθηκε το 2010 δεν προωθεί αρκετά το άρθρο 19 για την αυτόνομη ανεξάρτητη ζωή των ατόμων με αναπηρία. Ορισμένοι είχαν πει τότε ότι ήταν δύσκολο να προωθηθεί το άρθρο αυτό 19 και να ληφθούν σχετικές δράσεις. Νομίζουμε λοιπόν ότι μπορούμε εδώ πέρα να προωθήσουμε βέλτιστες πρακτικές για το άρθρο 19 και να καταφέρουμε να προχωρήσουμε και σε κάποια προγράμματα ευαισθητοποίησης. Έγινε ήδη μια συζήτηση για το ζήτημα της λιτότητας. Σας μας πει όμως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσο έχει πιέσει τα κράτη-μέλη προκειμένου να μην κάνουν δημοσιονομικές περικοπές όσον αφορά τα προγράμματα υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και πώς καταφέρνει να προωθήσει τελικά τις δράσεις για την αυτόνομη ζωή και την ένταξη στην αγορά εργασίας των ανθρώπων αυτών. Βλέπουμε ότι πολύ συχνά στα πλαίσια των πολιτικών λιτότητας είναι ακριβώς αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες υποχρηματοδοτούνται ή στις οποίες γίνονται περικοπές. Δράσεις δηλαδή, υπηρεσίες που έχουν ως στόχο να εντάξουν εκ νέου τα άτομα στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Και τέλος, όπως σας είπα, θα πρέπει τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δίνουν το καλύτερο θετικό παράδειγμα. Θέλουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς που να συμπεριλαμβάνει τα άτομα με αναπηρία, που θα χρησιμοποιεί τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα με τη συνεργασία του CRPD, όπου θα πρέπει να έχουμε την καλύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο όλοι από κοινού μπορούν να οδηγήσουμε σε μια καλύτερη διαβίωση των ανθρώπων αυτών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερχόμαστε τώρα στους εισηγητές και σκιώδες εισηγητές και επειδή πιέζει και ο χρόνος θα σας παρακαλούσα να περιοριστείτε σε ένα δίλεπτο. Όχι απλώς να το σκέφτεστε, να, προσανατολίζεστε, να το τηρείτε κιόλα. Η κυρία Χέλγκα Στέβεν, εισηγητή, έχει το λόγο. Γεια σας και ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ενδιαφερόμενους που απάντησαν στην πρόσκληση και ήρθαν ε, αυτοπροσώπως σε τόσο υψηλό επίπεδο. Αυτό δείχνει πόσο ψηλά είναι σε όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους ευρωβουλευτέ που ήρθαν και να σας δείξω ότι ε, Έχω εκπλαγεί θετικά και ευχάριστα από τον αριθμό των επιτροπών που γνωμοδοτούν. Δείχνει πόσο ενδιαφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα αυτό, τα μέλη. Επίσης, ε, είναι ένα θέμα οριζόντιο και εγκάρσιο και δεν μπορεί να περιοριστεί στα πλαίσια της δικής μας Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Παίζει ρόλο πρωταγωνιστικό και σε άλλες επιτροπές. Στο πνεύμα της σύμβασης Προσπάθησα ε, να έχω στενή συνεργασία με άτομα με αναπηρία και εκπροσώπους τους από ένα πρώιμο στάδιο για να είναι η έκθεσή μου και το έγγραφο εργασίας ε, όσο γίνεται πιο ε, πλήρες. Κάναμε και ακροάσεις και συνεδριάσεις του Intergroup ατόμων με αναπηρία, πάντα σε πολύ στενή συνεργασία, κυρίως με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αναπηρία και τα μέλη. Ίσως αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία στη σημερινή μας συνεδρίαση να πούμε ότι είναι από τις πιο προσβάσιμες συνεδριάσεις Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι σήμερα. Και θέλω να ευχαριστήσω τη γραμματεία της Επιτροπής για την πολύ σκληρή δουλειά και την υποστήριξη που μας παρήχαν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα έγγραφα εργασίας είναι πολύ σημαντικά, θέλω να τονίσω ορισμένα ζητήματα σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και πώς τα ίδια συμμορφώνονται προς τις ε, καταληκτικές παρατηρήσεις ε, του ΟΗΕ. Θα πρέπει εμεί να δίνουμε το θετικό παράδειγμα στα κράτη-μέλη και να βεβαιώσουμε ότι οι πολίτες μας, οι υπάλληλοι μας, αλλά και κάθε βουλευτής θα μπορούν να έχουν ε, απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις συνεδριάσεις και σε όλες τις εργασίες των θεσμικών οργάνων για τις δημόσιες συνεδριάσεις και ε, για τα όσα διοργανώνονται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως είναι η σημερινή συνεδρίαση. Συνάδελφοι, περιμένω τις απαντήσεις σας, περιμένω και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας και στη συνεργασία με τις άλλες επιτροπές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Άνταμ Κόζα τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Καταρχάς, θα ήθελα να καλωσορίσω τη σημερινή διοργάνωση, τη σημερινή συνεδρίαση. Χαίρομαι που ακούμε τις διάφορες οργανώσεις, τη διαμεσολαβήτρια, ε, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τους δύο εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών. Χαίρομαι για την ευκαιρία αυτή που έχουμε. Εδώ και χρόνια τονίζω αυτά τα ζητήματα. Και αυτό που είναι καλό για τα άτομα με αναπηρία είναι καλό για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Ο χάρτης αυτός δεν βοηθάει μόνο εμάς τους αναπήρους, αλλά και τους υπολείπους είναι καθημερινή δουλειά και καθημερινό πρόβλημα, ας πούμε, όταν κάποιος μιλάει γρήγορα και όχι μόνο όταν δεν μπορούν οι ανάπηροι να έχουν πρόσβαση σε ένα κτίριο ή ε, όταν δεν είναι ε, καλή η κατάσταση σε μια συνεδρίαση. Σας είπε και ο πρόεδρος ότι μια κυρία που κρατάει πρακτικά δεν είναι εδώ, είναι στο Αμβούργο και προβάλλονται στην οθόνη. Ε, Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν δουλεύεις σκεπτόμενος τους αναπήρους ε, βοηθάς και το γενικότερο πληθυσμό. Αυτό που με ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο και κατά πρώτο λόγο δεν είναι η έκθεση της κυρίας Στέβεν. Θέλω να μιλήσω λίγο για αυτά που ακούσαμε από τους εμπειρογνώμονες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχολείται συνεχώς ε, και με τα συμφέροντα των ατόμων με αναπηρία και το έχει κάνει. Είναι πάγιο αίτημα του Κοινοβουλίου. Είναι κρίμα που δεν ελήφθη υπόψη η γνώμη του ούτε συμμετείχε στη λήψη των αποφάσεων, γιατί το Κοινοβούλιο τα λέει αυτά ανέκαθεν. Όταν κυρώθηκε αυτή η σύμβαση, η συμφωνία, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκαναν μια διοργανική συμφωνία ε, αποκλείοντας το Κοινοβούλιο, το οποίο σήμερα καλείται να συμμετέχει. Τώρα, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο άκουσα μια παρατήρηση από τα Ηνωμένα Έθνη που λέει ότι οι τρεις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχουν και οι τρεις στην παρακολούθηση. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή την άποψη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό κοινοβούλιο παγκοσμίω όπου δεν έχουμε συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Ε, εκλεγόμαστε από το λαό άμεσα και γι' αυτό θα πρέπει να συμμετέχουμε και στον έλεγχο και στην παρακολούθηση. Εμείς δεν έχουμε δεσμεύσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε ε, είμαστε προσιλωμένοι προς τη μία ή την άλλη πολιτική κατεύθυνση. Κάτι που θέλω να τονίσω είναι το θέμα της ανεργίας. Είναι τραγική κατάσταση όπως καταλαβαίνετε. Και απασχόληση των αναπήρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 24% χαμηλότερη από το γενικό πληθυσμό. Χρειάζεται οπωσδήποτε βελτίωση. Και δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιούν τα άτομα με αναπηρία τα δικαιώματά τους. Το είπε και η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Ότι σε σύγκριση και σχέση με τον αριθμό των αναπήρων δεν έχουμε αρκετέ καταγγελίε και αρκετά παράπονα. Δεν το έχουν συνειδητοποιήσει και θα πρέπει να βοηθηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το πράξουν αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπλενκεβιτσούτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το εξαιρετικό αυτό έγγραφο εργασία. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι για πρώτη φορά έχουμε μία σφαιρική και εις βάθος συζήτηση με πάρα πολλούς αξιωματούχους από διάφορους φορείς. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε πλέον για την κατάσταση διαβίωσης των ατόμων με στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μία ανεξάρτητη παρακολούθηση της σύμβασης. Για ποιο λόγο. Έχουμε 28 κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η διαφορά από το ένα κράτος στο άλλο είναι πολύ μεγάλη. Η κατάσταση των ατόπων με αναπηρία στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφέρει επίσης πολύ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Η αντικειμενικότητα λοιπόν της παρακολούθησης θα μας επιτρέψει να δούμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία και μόνο κατά αυτόν τον αμερόληπτο τρόπο θα καταφέρουμε να λάβουμε αποφάσεις σε τοπικό, εθνικό και έπειτα ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, συμφωνώ ότι ε, θα πρέπει να αναφερθούμε και στη συνεργασία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε όμως να μιλάμε για μια ποιοτική τέτοια συνεργασία, μπορούμε να μιλάμε για μια επαρκή τέτοια συνεργασία, στον τομέα της ενσωμάτωσης και της ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Ας αποφύγουμε οποιαδήποτε αντιπαράθεση ή ανταγωνισμό ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επενδύσουμε περισσότερο σε μια ποιοτική συνεργασία με σωστικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι πρέπει εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο έγγραφό μας να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια ενδιάμεση αναθεώρηση τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία. Προφανώς στρατηγική αυτή που καλύπτει την περίοδο 2010 2020. Η εφαρμογή της σύμβασης αυτής, καθώς επίσης και να θεώρηση της σχετικής στρατηγικής, θα πρέπει να γίνουν από κοινού. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια αντικειμενική και πραγματική εικόνα της κατάστασης. Κάτι ακόμα. Απασχόληση των ατόμων με αναπηριακή ένταξή του στην αγορά εργασία. Η δική μα η Επιτροπή, η Επιτροπή Απασχόληση, πρέπει να μιλήσει για την πολύ δεινή κατάσταση που βιώνουν τα άτομα αυτά σε πάρα πολλέ χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την προσπάθειά του να ενταχθούν στην αγορά εργασία. Και κάτι ακόμα. Ξέρω ότι πολύ συχνά τα άτομα με αναπηρία δεν έχουν τα απαραίτητα κίνητρα για να ενταχθούν στην αγορά εργασία και αναφέρομαι βέβαια σε μια ανοιχτή αγορά εργασίας και όχι μόνο σε μια περιχαρακωμένη αγορά εργασίας που να προορίζεται μόνο για αυτούς συγκεκριμένα εργαστήρια για παράδειγμα τα οποία αποφασίζουν να τους δώσουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν στην ατομέα. Και κάτι ακόμα. Ας μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια ελάχιστα πρότυπα κοινωνικής προστασίας για τα άτομα με αναπηρία. Ας μην ξεχνάμε ότι ε, τα άτομα αυτά δέχονται πρώτα από όλου και περισσότερο από όλου τις ε, δεινές συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Είμαι επίσης σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς επίσης και με άλλους σχετικούς φορείς εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να ακούμε πρώτα τη δική τους τη φωνή, προτού τοποθετηθούμε εμείς με τον ένα τον άλλο τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ όμως να τηρείτε τον χρόνο ομιλίας. Η κυρία Χάρκιν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα περιοριστώ στο δίλεπτο. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές μας σήμερα το πρωί. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμες οι παρεμβάσεις σας και νομίζω ότι μας ε, δώσατε ένα πλαίσιο εντός του οποίου μπορούμε να κινηθούμε. Επίσης χάρηκα που μπόρεσα να συμμετέχω σε μια συνεδρίαση με πραγματική προσβασιμότητα και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους οργάνωσαν την συνάντηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Χέλγα Στίβενσε για το εξαιρετικό της το οποίο νομίζω ότι παρέχει ένα καλό πλαίσιο εντός του οποίου μπορούμε να εργαστούμε. Δεδομένου του περιορισμένου μου χρόνου, θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Ε, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να απαντήσουν, αλλά θα θέσω τις ερωτήσεις μου. Η Diane Kingston αναφέρθηκε στα προστατευμένα εργαστήρια. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το επόμενο βήμα. Θα ήθελα όμως να ακούσω τις απόψεις σας, διότι και ο συνάδελφος ε, από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, μίλησε για πραγματικές θέσεις εργασίας και όχι προστατευμένες θέσεις εργασίας. Και Μήπως μπορείτε να μας δώσετε ιδέες σχετικά με το πώς μπορούμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Όχι απαραίτητα με νομοθεσία, αλλά ε, με κατευθυντήριες γραμμές, ε, με προγράμματα μεντόρων. Ε, πώς μπορούμε να προοδεύσουμε στον τομέα αυτόν. Ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε σήμερα το πρωί από αρκετούς από τους ομιλητές ήταν το θέμα της λιτότητας. Και Αυτό σχετίζεται και με το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Πολλοί μίλησαν για, τη, για τις ανάλογες επιπτώσεις ε, της λιτότητας ε, στα άτομα με αναπηρίες ε, και ζητήθηκε να μην γίνουν περικοπές ιδιαίτερα για την αυτόνομη διαβίωση και τις σχετικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο λοιπόν του Ευρωπαϊκού εξαμινού, μπορούμε να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ιδιαίτερα στις συστάσεις αναχώρα να συμπεριλαμβάνει τέτοιες συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Ε, ναι, ξέρω, είπα ότι θα μιλήσω από δύο λεπτά, δέκα δευτερόλεπτα δώστε μου ακόμα. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια ε, διαβούλευση μέχρι τον Μάρτιο του 2017. Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι σχετικοί οργανισμοί να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή για να λάβουμε υπόψη μας τις παρατηρήσεις τους ε, κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση της ε, πράξης για τα άτομα με Σε Ευχαριστώ. Ε, σε ευχαριστώ Μάρια. Ναι, ε, ναι, οι καλές σου προθέσεις φάνηκαν πάντως. Ε, το λόγο έχει η Κωνσταντίνικα Κακούνεβα. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και σε όλους που ήρθαν σήμερα και συζητήσαμε επάνω στο θέμα. Ευχαριστώ και εγώ την Μιχαήλ Στίβεν για την δουλειά που κάνει για αυτή την τόσο σημαντική για την κοινωνία μας έκθεση διαβάζοντα το ιστορικό τη σύμβαση του ΟΕΕ, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, καθώ και το έγγραφο εργασία που μα παρουσίασε η συνάδελφο Χέλεγα Στίβαν, διαπιστώνουμε κάτι παράδοξο. Πέντε χρόνια από τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά ω εννέα οντότητα προσχώρησε στη Διεθνή Σύμβαση, διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να την εφαρμόζει στο σύνολό τη. Γιατί διότι ανακαλύπτει καθυστερημένα ότι πολλές από τις επιταγέ της σύμβασης είναι η εθνική αρμοδιότητα των κρατών μελών και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σύνολο. Αυτό το θεσμικό έλλειμμα είναι υπαρκτό. Αλλά νομίζω ότι χρηματο... χρησιμοποιείται από την Κομισιόν και σαν πρόσχημα. Τόσο η Κομισιόν όσο και το Συμβούλιο θυμούνται επιλεκτικά πότε έχουν πότε έχουμε γενοσιακό δίκαιο και πότε ένα θέμα είναι υποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όταν όμω εφαρμόζουν του κοινού κανόνε τη δημοσιονομική λιτότητα που επιχειρεί, επηρεάζουν κάθε πεδίο πολιτική, είτε είναι εθνική είτε ευρωπαϊκή, είναι πάντα αυστηρή και άκαμπτη και αδιάφοροι για το τι επιπτώσεις έχει η λιτότητα και στα άτομα με αναπηρία. Αντίθετα τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχεται από την Επιτροπή Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ότι δεν εφαρμόζει με συνέπετο τη σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων η Κομισιόν λέω ότι τα χέρια της είναι δεμένα. Οχυρώνεται πάλι πίσω στην φράση «εθνική αρμοδιότητα». Νομίζω ότι η σύμβαση του ΟΕΕ και τα προβλήματα εφαρμογής της είναι μια ακόμα ευκαιρία για να αναδείξουμε ένα ζήτημα τεράστια πολιτική σημασία για την επιβίωση τη ίδια τη Ευρώπη. Είναι απλό. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να αποκουτεύσει για άλλη μια φορά του πολίτε τη, όπω έχει συμβεί συχνά τα τελευταία χρόνια, οφείλει να υιοθετήσει κοινέ πολιτικέ σε τόσο ευαίσθητα ζητήματα πρέπει να θεσμοποιήσει αυτές τις πολιτικές. Ακόμα και αν χρειάζονται αλλαγές τι συνθήκε, οι νέα νομοθετήματα και νέοι πόροι χρηματοδότηση. Μακάρι η πλήρη εφαρμογή στι συμβάσει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία να είναι εφαρμογή για ένα ακόμα βήμα για περισσότερο Ενωμένη Ευρώπη. Επομένω, νομίζω ότι η έκθεση που τα εγκριτεί η Επιτροπή μα πρέπει να απαιτηθεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που βρίσκονται εκτός ενωσιακής πολιτικής. Δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικίνητρο για δράση, αλλά κίνητρο για να διαμορφώσουμε τα αναγκαία παιδεία κοινή πολιτική. Δεν είναι θέμα αξιοπρέπειας των αναπήρων, είναι θέμα αξιοπρέπειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Τατιάνα Στάνοκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την Χέλκα Στίβενς για την δουλειά που ήδη έχει κάνει σε προετοιμασία της έκθεσης αυτής. Έχει συνεργαστεί στενά με μη κυβερνικές οργανώσεις έχει οργανώσει συναντήσεις με μη οργανώσεις, στις οποίες συμμετείχα και εγώ. Θα ήθελα να αδράξω και την ευκαιρία να καλωσορίσω τον συμπατριώτησα μου Γκούντα Άνκα που συμμετέχει στη σημερινή συζήτηση. Θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην Χέλγα στις ε, περαιτέρω εργασίες πάνω στην έκθεση αυτή. Θα υποβάλουμε φυσικά τις προτάσεις μας. Ε, τώρα όμως ε, στην πρώτη συζήτηση σημαντικό είναι η εφαρμογή της ε, σύμβασης του ΟΗΕ να ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτομα με αναπηρίες. Είναι σημαντικό λοιπόν να συνδυαστήμες εργασίες πάνω στην ε, οριζόντια οδηγία, ε, θέμα που παραμένει προβληματικό. Σημαντικό είναι επίσης εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης ε, να ασχοληθούμε και με το θέμα απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες. Και το θέμα δεν είναι να προσαρμοστούν αυτοί στην υπάρχουσα αγορά εργασίας, αλλά να εξετάσουμε γενικά την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να προσαρμοστεί η αγορά εργασίας στις δικές τους δυνατότητες και ικανότητες. Είναι επίσης σημαντικό να εντατικοποιηθούν οι εργασίες ε, κατά τις... Ε, Τοποθέτηση των ανθρώπων ε, σε ιδρύματα ιδιαίτερα. στις περιπτώσεις ε, νέων και παιδιών με αναπηρίες. Δεν πρέπει να τους αποκλείσουμε από την κοινωνία μας, θα πρέπει να τους ανοίξουμε την πόρτα. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες κύριες ιδέες και φυσικά γνωρίζουμε ότι δεν έχουν εφαρμόσει όλα τα κράτη-μέλη αυτήν την σύμβαση. Ελπίζω Ελπίζω η εξέταση και των 28 κρατών μελών ε, σχετικά με το πού βρίσκονται όσον αφορά την εφαρμογή της σύμβασης να συμπεριληφθεί στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η Λαουρά Ατζέα. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε και καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο υποδέχεται μια σημαντικότατη συζήτηση σήμερα και πάρα πολλούς σημαντικούς αξιωματούχους και φορείς. Το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και οφείλουμε εμείς να συμβάλλουμε κατά τρόπο αποτελεσματικό. Δυστυχώς, συντοποιούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο από ότι η δική μου η χώρα. Έννοιες όπως η αποδρυματοποίηση, η ένταξη των ατόμων στην αγορά εργασίας απέχει πάρα πολύ από το να αποτελούν πραγματικότητα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όντως να γίνει αυτή η εργασία παρακολούθησης όπως είπε και μια συνάδελφος πριν από λίγο για να βλέπουμε πραγματικά πώς εφαρμόζεται η σύμβαση αυτή στα κράτη-μέλη τα ίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί τελικά να βλέπει πώς εντάσσονται ή όχι τα άτομα με αναπηρία στην κοινωνία, στην αγορά εργασίας. Εμείς κάνουμε πάρα πολλά αιτήματα μέσω της ε, έκθεσής μας αυτής, πράγμα το οποίο δείχνει ότι όντως υπάρχουν πάρα πολλά κενά ακόμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε ποια είναι η ίδια η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ίδια η στάση των κρατών μελών της Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο θα πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε για τα ζητήματα αυτά, να συζητάμε για τα ζητήματα αυτά, να πετούμε περισσότερη ενσωμάτωση στην ατόμων αναπηρία στις κοινωνίες μας. Εγώ θα ήθελα άνθρωποι όπως ο ανιψιός μου ή πολλοί άλλοι γνωστοί μου και φίλοι να μπορούν πραγματικά να ενηλικιωθούν σε έναν κόσμο φιλόξενο, σε έναν κόσμο που πραγματικά θα είναι σε θέση να τους υποδεχθεί. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και ιδιαίτερα που τηρήσατε το δίλεπτο. Ζωέλ Μεράν, παρακαλώ. Ε, euh, euh, euh. Ευχαριστήσω καταρχάς την εισηγήτρια την κυρία Στίβεν, η οποία επικεντρώθηκε στα ζητήματα εκείνα τα οποία τονίζονται περισσότερο στις τελικέ παρατηρήσει. Αναφέρεται όντω εδώ πέρα στι συστάσει, οι οποίε αντιστοιχούν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκή Ένωσης και οι οποίες δημιουργούν κάποια προβλήματα κατά την εφαρμογή του στα κράτη-μέλη. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε νομοθετικές πράξεις οι οποίες έχουν ευρωπαϊκό καθαρά χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα η οδηγία για την διασυνοριακή παροχή υγειονομικών υπηρεσιών ή την οδηγία για την ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση ή την οδηγία για την ισότιμη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η κυρία Στίβεν αναφέρθηκε στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα ίδια τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούν να δώσουν το θετικό παράδειγμα για την εφαρμογή τη σύμβαση αυτή. Αναφέρθηκε σε ζητήματα όπω οι συνθήκε απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κανονισμό υπηρεσιακή κατάσταση κ.ο.κ η κυρία Στίβενς θεωρεί ότι δεν προβλέπεται εδώ πέρα κάποια ιεράρχηση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι η διάκριση η οποία βασίζεται στην αναπηρία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η διάκριση ή διακρίσεις για άλλους λόγους, όπως για παράδειγμα οι πολλαπλές διακρίσεις. Η διακρισει για αλλους λογους αυτή είναι πολύ σημαντική και αφορά κυρίως τις γυναίκες και τα παιδιά τα οποία πλήττονται και από αναπηρίες. Ιδίως όσον αφορά επίσης την ε, νοητική υστέρηση, τις ε, ψυχοκοινωνικές αναπηρίες. Τα ζητήματα αυτά μας αφορούν όλους ιδιαιτέρως. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της σύμβασης αυτής. Και ολοκλήρω την παρέμβασή μου σε 1 λεπτό 44 δευτερόλεπτα, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ που τηρήσατε και τον χρόνο. Έχουμε πέντε ομιλητές στον κατάλογο, από ένα λεπτό ο καθένας. Ένα λεπτό. Εάν ε, δεν τηρήσετε το χρόνο θα ε, βάλω διακόπτη ώστε να μπορώ να κλείνω το διακόπτη. Α, υπάρχει τέτοιο διακόπτη. Ήδη, ωραία. Μπενιφέη, παρακαλώ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την κυρία Στίβενς γιατί πραγματικά θέτει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ζήτημα αυτό. Ο χρόνος πιέζει θα είμαι πολύ σύντομος και άμεσος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δική μας την έκθεση του Κοινοβουλίου να περιλάβουμε τέσσερα ζητήματα ανεξάρτητο πλαίσιο παρακολούθησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, διοργανική επίσης συνεργασία μεταξύ Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπόλοιπων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να έχουμε μια νέα θεσμική ευτεκτονική όσον αφορά την πολιτική για τα άτομα αναπηρία. Νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να βαθώνουμε περισσότερο για το πώς το ευρωπαϊκό εξάμεινο θα μπορούσε να συμβάλλει στην εφαρμογή της σύμβασης αυτής τρίτων, αναθεώρηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα άτομα αναπηρία, προκειμένου η στρατηγική αυτή να είναι σφαιρική, ολιστική και τέταρτο και τελευταίο σημείο, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια ολοκληρωτική αναθεώρηση της κοινοτικής νομοθεσίας, προκειμένου να συνάδει περισσότερο με την σύμβαση. Επί των σημείων αυτών είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με όλους τους συναδέλφους και να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την εισηγήτρια. Δίτερ κόχ παρακαλώ ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και χαίρομαι που θα υπάρξει έκθεση πρωτοβουλίας. Θα πρέπει να υπάρχει χώρος για όλους στην κοινωνία μας και ιδιαίτερα των 80 εκατομμυρίων ανθρώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που έχουν ε, αναπηρίες. Ε, η ζωή τους εμποδίζει. Θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να έχουν πρόσβαση σε παιδεία, περίθαλψη υγείας, κοινωνική προστασία μέσα μαζικής μεταφοράς ε, και πληροφορίες. Είμαι ευγνώμων ε, στην εισηγήτρια. που αναφέρθηκε και στον ε, αριθμό κλήσης για επίγοντα 112 που θα είναι κοινός για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρω ότι περιμένετε την ε, ψηφοφορία, αλλά μήπως μπορείτε να κάνετε λίγο περισσότερη ησυχία. Λάμπρος Φουντούλης, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα σήμερα να μιλήσω πρώτα σαν πατέρα μια κόρη με ειδικέ ανάγκε και μετά σαν Ευρωβουλευτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Στίβεν, για τη δουλειά τη. Δυστυχώ σε όλε τι χώρε τη Ένωση τα άτομα με αναπηρία δεν έχουν τι ίδιε ευκαιρίε και την ίδια ποιότητα ζωή όπω θα έπρεπε. Θα μιλήσω για τη χώρα μου, την Ελλάδα. Τα άτομα με αναπηρίε και οι οικογένειέ του είναι τα μεγαλύτερα θύματα τη οικονομική κρίση. Στο πλαίσιο τη δημοσιονομική προσαρμογή στην Ελλάδα έχουν γίνει περικοπέ μισθών και συντάξεων στου γονεί των παιδιών με αναπηρία. Πώ μπορούν να προσφέρουν οι γονεί αυτοί τα απαραίτητα στα παιδιά του για αξιοπρεπή διαβίωση και τι αυξημένε ανάγκε που έχουν τα άτομα με αναπηρία σε σχέση με του άλλου συνανθρώπου μα. Η αυτόνομη διαβίωση στην Ελλάδα δεν υπάρχει με τη μέρημνα του κράτου. Μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει κάνει κάποια βήματα στον τομέα αυτό, αλλά αντιμετωπίζεται σαν επιχειρηματία και εξοντώνεται με υπέρμετρη φορολόγηση. Τα άτομα με αναπηρία έχουν εξαιρεθεί από τα προγράμματα διαβίου μάθηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ακόμα και απλά θέματα όπω είναι μια θέση πάρκινγκ έξω από την κατοικία των ατόμων αυτών δίδεται μόνο αν έχουν τα ίδια τα άτομα δικό του αυτοκίνητο. Πρέπει όλοι να έχουμε μια ενιαία στάση υπέρ των δικαιωμάτων των συνανθρώπων μας με αναπηρία, γιατί οι ανάγκες είναι καθημερινές και κοινέ για όλους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Χέλκα Στίβενς και όσου συμμετέχουν στον επικοδομητικό διάλογο για ε, τη σύμβαση των ατόμων με ειδικέ ανάγκε. Θα ήθελα να επισημάνω κάτι σημαντικό όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των ε, ατόμων με αναπηρίες. Αναφέρομαι στους κοφούς. Λίγα κράτη-μέλη παρέχουν σε χρήστες της νοηματικής την δυνατότητα διερμηνία στις επαφές με τις αρχές. Αυτό δεν παρέχεται πάντα και έτσι δεν διασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων που χρειάζονται τέτοια βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και έχουμε τώρα τον τελευταίο μιλητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι γνωστό ότι η στάση που έχουμε απέναντι στα άτομα με αναπηρία δείχνει τελικά και για κάθε χώρα πόσο προηγμένη είναι ή πόσο προηγμένη δεν είναι. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να παρέχουμε ισότιμη μεταχείριση σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα με το αν πλήττονται από κάποια αναπηρία ή όχι. Βλέπω παρόλα αυτά ότι υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον συνδυασμό των διαφορετικών απόψεων που έχουν ακουστεί όσον αφορά την ένταξη των ανθρώπων αυτών στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Αναφερθήκαμε σε πραγματικές θέσει απασχόλησης, σε πραγματικές επιχειρήσει και εταιρείε. και να γίνει κάτι τέτοιο, χρειαζόμαστε συγκεκριμένη ευρωπαϊκή στρατηγική. Ευχαριστώ. Τώρα θα παρακαλέσω τους εμπειρογνώμονες να απαντήσουν. Ένα λεπτό έκαστος γιατί δεν έχουμε χρόνο. Στις ερωτήσεις παρακαλώ να απαντήσετε μόνο. Τώρα έχω χάσει και τη σειρά. Θέλω να μιλήσουν όλοι. Ε? Η Ντάιν Κίνγκστον πρώτη. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καταπληκτικές αυτές ερωτήσεις και τις παρεμβάσεις σας. Να απαντήσω σε δύο παρεμβάσεις. Πρώτον, όσον αφορά τα εργαστήρια αυτά, τα περιορισμένα, περιχαρακωμένα, οριοθετημένα που προορίζονται για τα άτομα αναπηρία, καθώς επίσης και τα όσοι υπόθηκαν για την αποϊδρυματοποίηση. Νομίζω ότι η αποϊδρυματοποίηση και ένταξη στην αγορά εργασίας μπορεί να γίνουν παράλληλα. Αναφερθήκατε επίσης κατευθυντήρες γραμμές βελτίστων πρακτικών για την ένταξη των ανθρώπων αυτών στην αγορά εργασίας. Αναφερόμαστε εδώ πέρα στη δυνατότητα πρόσληψης, διατήρησης και προώθησης προαγωγής των ανθρώπων αυτών στα πλαίσια μιας εταιρείας. Η στην υπαριθμόν 2 παρατήρηση, καταληκτική παρατήρηση των ΗΕ μπορείτε να δείτε σχετικές ε, μνήες που γίνονται για την προσβασιμότητα αυτή και μπορώ να σας δώσω βέβαια εγώ και περισσότερες πληροφορίες για το ζήτημα αυτό. Δεύτερον, να απαντήσω στον Άνταμ Κόσα. Όσον αφορά το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την παρακολούθηση τη εφαρμογή τη Σύμβαση των Ηνωμένων και ως προς αυτό να πω κάτι πολύ σημαντικό. Η εφαρμογή της σύμβασης και η παρακολούθηση της εφαρμογής σύμβασης είναι δύο ξεχωριστές αρμοδιότητες, δύο ξεχωριστοί ρόλοι που δεν θα πρέπει να επικαλύπτονται. Η παρακολούθηση θα πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητη. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμπλέκεται στην εφαρμογή της σύμβασης, δεν μπορεί να εμπλέκεται και στην παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης. Επ' αυτού μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες μέσω των αρχών των Παρισίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μάικλ Φλάχερτη. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω σήμερα στην ερώτηση που τέθηκε της κυρίας Χάκνη σχετικά με τα ιδρύματα. Ας σταματήσουμε να στηρίζουμε οικονομικά τα ιδρύματα με ε, πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρει η Κομισιόν ε, στα συμπεράσματα. Και επίσης, Ας ε, υιοθετήσουμε την ε, σύσταση του EDF ε, καθώς και την παράγραφο 71 που ζητεί επικύρωση της σύμβασης του Μαρακές. Και τρίτον, να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία της του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να χρησιμοποιηθούν και στην διαμόρφωση πολιτικής και νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Η Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα νομίζω ότι ακούστηκαν ε, διάφορες παρατηρήσεις. Ε, δεν μπορώ να σχολιάσω όλα όσα υπόθηκαν, αλλά σίγουρα χρειάζεται να γίνει συζήτηση όσον αφορά ε, την ανεξαρτησία της, του πλαισίου παρακολούθησης. Σίγουρα πολύ. Ε, ενδιαφέρονται για την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων ε, όσον αφορά όχι τη σύμβαση αλλά γενικά την ε, κατάσταση ανθρώπων με αναπηρίες. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα δυναμική. Υπάρχει μια αίσθηση στασιμότητας, χρειαζόμαστε κυρίως πολιτικούς που θα προβάλλουν τα θέματα αυτά. Φυσικά ε, θα πρέπει να αποφεύγουμε την ε, ιδρυματοποίηση, και αυτό ε, ιδιαίτερα εδώ την τελευταία ώρα και έχω εξετάσει το θέμα αυτό σε σχέση με το πώς δαπανώνται οι πόροι του Ταμείου Συνοχής και το πώς δαπανούν τα κράτη-μέλη του πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κούντα Άνκα. Ευχαριστώ πολύ και να σας ευχαριστήσω για τις καταπληκτικές αυτές παρατηρήσεις και παρεμβάσεις που άκουσα σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είδα ότι ε, εμπλέκονται αρκετοί ευρωβουλευτές στο ζήτημα αυτό, αλλά έχουμε και βουλευτές πολλές φορές ε, εκτός κοινοβουλίου που ενδιαφέρονται πολύ. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα χωρίς την εμπλοκή των ανθρώπων με αναπηρία. Είναι σημαντικό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία να εμπλέκεται. Εθνικοί φορεί εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία επίση πρέπει να εμπλακούν και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να οδηγηθούμε σε θετικά αποτελέσματα ουσιαστικά και όχι μόνο σε θετικέ εκθέσει. Σήμερα μιλήσαμε πάρα πολύ για το ζήτημα της απασχόλησης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να έχουμε μια ανοιχτή αγορά εργασίας για τα άτομα αναπηρία. Τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά βέβαια. Πρέπει να δούμε τι υποστήριξη μπορούμε να παράσχουμε στους ανθρώπους με αναπηρία, προκειμένου να μπορούν να εισέρχονται και να παραμένουν σε μια ανοιχτή αγορά εργασίας. Η υποστήριξη χρειαζόμαστε σε πάρα πολλούς τομείς μόνο, όχι μόνο στον τομέα της απασχόλησης. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν και τους άλλους κλάδους. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο Γιάννη Γιάραπ. Ευχαριστώ όσον αφορά το ζήτημα της αποεδρυματοποίησης. Να σε επαναλάβω ότι έχουμε ένα έγγραφο Ευρωπαϊκές Κατευθύνες Γραμμές για τη μετάβαση από τα Ιδρύματα στην κοινωνία που δημιουργήθηκε από το συνασπισμό αυτό που, αναφέρθηκα πριν από λίγο, που ανέφερα πριν από λίγο, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει μεταφραστεί ήδη σε αρκετέ γλώσσε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχετικά σεμινάρια γίνανε επίση για το ζήτημα αυτό. 14 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν συμμετάσχει και έχει ξεκινήσει μια σχετική διαδικασία σε πολλέ από τι χώρε αυτέ. Α μιλάμε λοιπόν, δεν έχει συμβεί τίποτα για το ζήτημα αυτό. Ήδη από το 2010 και μετά, πολλά κράτη-μέλη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν το έγγραφο αυτό, τι κατευθυντήρε αυτέ γραμμέ, προκειμένου να σημειώσουν πρόοδο στη διαδικασία αυτή της αποϊδρυματοποίησης. Όσον αφορά το ζήτημα της απασχόλησης, ένα ερώτημα που ετέθη είναι πώς μπορούν τα άτομα με αναπηρία να ενταχθούν σε μια ανοιχτή αγορά εργασίας και όλοι μας είπαμε ότι το εγχείρημα αυτό είναι σίγουρα δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά έχουμε ήδη κάποια θετικά ενθαρρυντικά παραδείγματα μέσω των προγραμμάτων αυτών ε, απασχόλησης με την παροχή υποστήριξης όπου προσπαθούμε να έχουμε καταρχάς μια σωστή κατάρτιση, καθοδήγηση στην ατόμο αναπηρία και να υπάρχει στη συνέχεια μια καλύτερη αντιστοιχία ανάμεσα στις δεξιότητές τους και τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης. Νομίζω ότι τα παραδείγματα τα οποία είχαμε μέχρι στιγμής ήταν θετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συγγήτρια θέλει ξανά το λόγο. Έχετε τη δυνατότητα κυρία Στέβεντς να ξαναμιλήσετε αν θέλετε. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη επειδή δεν έχουμε χρόνο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους, ιδιαίτερα όλους τους συναδέλφους, ευρωβουλευτές, συν όλους τους υπόλοιπους που ήρθαν από οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όργανα παρακολούθησης, ε, φορείς αναπήρων. Σας ευχαριστώ όλους για τη μόνιμη και πάγια εισφορά σας και θέλω στο μέλλον ε, να συνεχίσετε να μας βοηθάτε, να ακούμε τα σχόλιά σας και τα λοιπά. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ εμπεριστατωμένη η συζήτηση. Από χρόνο δεν πάμε πολύ καλά. Ένα σύντομο σχόλιο στο τέλος. Δεν έχουμε μπει ακόμα σε θέματα εφαρμογής ούτε καν ελέγχου. Αυτή τη στιγμή ακόμα είμαστε στην πρωτοβουλία της Επιτροπής μας ε, για να στηθεί αυτή η προσπάθεια, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εργαζόμαστε πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολύ ε, προσιλωμένοι σε αυτή την υπόθεση για να ε, προκύψουν κάποιες ρυθμίσεις βιώσιμες. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες, τους ομιλητές και ε, τις διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας, αλλά και τους δικούς μας διερμηνείς της καμπίνες ήταν κάπως δύσκολη η σημερινή αφετηρία και η κίνηση από τεχνική πλευρά. Ευχαριστώ και την κυρία Στομβούργο που τα γράφει όλα αυτά, αλλά και την γραμματεία που έχει κάνει τρομερή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ για τη διοργάνωση αυτή. Θα διακόψουμε εδώ για να πάμε στο επόμενο θέμα που είναι οι ψηφοφορίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στο σημείο 5 τη ημερήσια διάταξης που είναι έγκριση γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίηση. Äh, είναι η περίπτωση ενώ να μην γκλάς Βέλγιο. Εισηγητής, α, εγώ είμαι μάλλον, εντάξει. Όλα καλά. Είναι μία και μοναδική ψηφοφορία εδώ, ηλεκτρονικά. Παρακαλώ να ψηφίσουμε για το σημείο 5, ε, υπέρ έρχεται η ψηφοφορία. Η Abstimmung ist eröffnet. Τώρα αρχίζει. Oh, Εγκρίθηκε, αλλά από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα περισσεύουν δύο και από τους σοσιαλιστές ένας υπεράριθμος. Ντέιβιτ και Γιούτα, μπορείτε να το λύσετε παρακαλώ πολύ οι ε, συντονιστές. Ακόμα ένας υπεράριθμος από τους σοσιαλιστές, το ΕΛΚ είναι εντάξει. Τώρα είμαστε όλοι εντάξει, ωραία, αλλά πρέπει να ξαναψηφίσουμε γιατί περίσσευαν τρει προηγουμένω τώρα ξαναρχίζει η ψηφοφορία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο παγκοσμιοποίηση στο σημείο 5. Πάλι ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ. David Κάζα, μπορείτε λίγο να το ρυθμίσετε εκεί τις γραμμές του ΕΛΚ. Τώρα εντάξει. Λοιπόν, 47-6 τώρα εγκρίνεται επίσημα και κανονικά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο σημείο 6, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών κλπ. Η συγκήτρια είναι η κυρία Σοφία Ριβέιρο. Είναι αρκετά χοντρή ψηφοφορία τώρα αυτή που έχουμε μπροστά μας. 430 συνολικά τροπολογίες. 6 τροπολογίες για το gender mainstreaming και 57 παρακαλώ συμβιβασμοί που φιλοδοξούν και προσπαθούν να καλύψουν αρκετά πράγματα αλλά όχι όλα. Πάμε λοιπόν. Η τροπολογία 121. Η πρώτη. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική S-α. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική S. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα που πάμε έχουμε και τα χρωματάκια μας εδώ. Compromise T. Συμβιβαστική T υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική V υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 160 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε, X υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά 167 το δεύτερο τμήμα ω συμπλήρωση της συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε συμβαστική Z, Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 182 ψήφι υπέρ κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία, είμαστε στην τροπολογία 182. Πάλι ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ. Εξακολουθεί. David Κάζα. Μην κάνεις τέτοιους μορφασμούς, σε παρακαλώ. Ξανά. Ψηφίζουμε την 182 τροπολογία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Και με μεγάλη διαφορά. Ε, συμβαστική ΑΑ υπέρ. Κατά. Απόχε, εγκρίνεται. Η 188 υπέρ. Κατά. άποχέ. Απορρίπτεται 189 υπέρ. Κατά. Απόχε. Απορρίπτεται. Συμβαστική ΑΑΒ μικρό υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 286 έχει αποσυρθεί και πάμε στο συμβιβασμό ΑΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 208 υπέρ κατά Απόχες εγκρίνεται. Συμβαστική ε, AC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 212 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Ας το ελέγξουμε αυτό παρακαλώ. 212 ελέγχουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 25-24. Με μικρή διαφορά εγκρίθηκε. 213. είπε. Κατά. Και αυτό θέλει έλεγχο. Γιατί δεν βλέπω τι ψηφίζεται και τι δίνουν τα WIP. Τη 213 ψηφίζουμε. Αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίφτεται. Ωραία. Συμβαστική αντέ είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική αντέ αλφα μικρό είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική εψιλον, είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 232 ψήφι Πέ, κατά αυτό θέλει έλεγχο. Η 232 επαληθεύεται ηλεκτρονικά, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Πάμε στη 233 ψηφίπε. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 233 Αρχής τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 234 υπέρ κατά αποχές έλεγχος με τη 234. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία και κλείνει αμέσω. Εγκρίθηκε. 235 είπε. κατά αποχές έλεγχος και για τη 235 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Ορίστε. Έτοιμοι. Καλώς. Έχετε τίποτα θέματα να συζητήσετε, να λύσετε. Όχι. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίθηκε 30-23. Είμαστε τώρα στη 236 ψήφι πέρα. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΕΦ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα είμαστε στην τροπολογία μισό να τη βρω 251. Έτσι δεν είναι είπε. κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ήτα είπε. κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολόγια 252 είπε. Όχι, συγγνώμη, έχει αποσυρθεί λέει ο πρόεδρος. Ναι, δεν το διάβασα. Συμβαστική ΑΓ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΙ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 271 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 272 υπέρ κατά αποχές αυτό απορρίπτεται μάλλον. Απορρίπτεται. 273 υπέ. Κατά αποχές. Και αυτό απορρίπτεται. Τσεκ. Καλά, ας το ελέγξουμε. Την 273 λέει ο Πρόεδρος. Ψηφίσατε όλοι. Τέρας. 25-23 εγκρίνεται. Sorry. 274 είπε Κατά. Γεια σας. Αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική ΑΚ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΛ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 289 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 291 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 292 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 293 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ε, αλφαμή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 302 έχει αποσυρθεί, 303 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος για την 303. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. abgestimmt, Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. 304 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφτεται. Συμβαστική α, μη α μικρό υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Η 309 υπέρ όχι. Περάσαμε μια συμβιβαστική. Α, πολύ τρέχω σήμερα. Λοιπόν, συμβαστική αλφανή είναι αυτή τότε. Έτσι, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 309 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική αλφαόμικρον υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική αλφαπή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά έχουμε την 326 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 327 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίψεται. Συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΕΣ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΤΑΦ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΙΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ...344 τώρα, με μια προφορική τροποποίηση που βλέπετε εδώ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΒ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική w, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική w, α μικρό υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 357 έχει αποσυρθεί συμβιβαστική ΑΧ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 366 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, Συμβαστική ΑΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η συμβαστική ΑΖ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 382 υπέρ Α, όχι, συγγνώμη, έχουμε κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, είπε Κατά. Αποχές. Έλεγχος, γιατί δεν είναι σαφές, 382 το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Και αν ψηφίσατε όλοι, πέρασε. Απορρίφτεται. Το δεύτερο τμήμα πρέπει να το ψηφίσουμε. Mm? Πρέπει μάλλον, ε. Άρα ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ορίστε. Συμβαστική ΒΑ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΒΑ κεφάλαιο α μικρό. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β, α κεφαλαίο Β μικρό, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η, τώρα, η 395 ψήφι Π, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 396 υπέρ, κατά, αυτό δεν το κατάλαβα. Παρακαλώ να την ελέγξουμε. 396 ηλεκτρονική απορρίθωση. Αν ψηφίσατε όλοι κλείνει. Απορρίπτεται. 397 υπέ, κατά αποχές. Νομίζω η ίδια αλλά για καλό και για κακό το ψηφίζουμε 397 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Φέρες. Α, εγκρίθηκε. Ω. Τρία υπέρ. Υπέρ κατά αποχές. Δεν είναι πολύ σαφή τα πράγματα και εδώ χρειάζεται έλεγχο. Είναι μοιρασμένα. 398 ψηφίσμοι ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πιο αφές αυτό. Έπρεπε να το είχα δει. Απορρίπτεται. Συμβαστική ΒΒ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. τα έχουμε την 300 όχι έχουν καταπέσει αυτά, 403 είναι το επόμενο υπέρ, κατά αποχές απορρίψετε, δηλαδή εγκρίνεται, διορθώνει ο πρόεδρος, ζητά και συγγνώμη, 403 εγκρίθηκε για τα πρακτικά, 404 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 405 υπέρ, κατά απορρίψετε, συμβαστική ΒΒ σι μικρό, υπέρ, κατά άποχες εγκρίνεται συμβαστική β, β, α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 415 υπέρ κατά απορρίψεται Συμβαστική βήταση. Τσεκ, πολύ ωραία. Ελέγχουμε τη 415, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρα. Τι έχουμε εδώ. Απορρίπτεται. Καμιά φορά το πιάνω κιόλα. Ε, συμβαστική εμπίση Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 423 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβαστική BD υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται συμβαστική ΒΕ ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στις αιτιολογικές αναφορές τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται, τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, η τροπολογία 8 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται, η τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 13 καταπίπτει 28 και 30 όλα αυτά καταπίπτουν και πάμε στην 11 μάλλον Είμαστε στην 11. Συμφωνείτε. Ωραία. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 14 έχει καταπέσει. Και 25. Και πάμε στη 15 τώρα. Τροπολογία ψήφι υπέρ. Κατά αποχές. Τώρα αυτό θέλει έλεγχο παρακαλώ για την τροπολογία 15. Ψηφίσατε όλοι, πέρας μην Η τροπολογία 16 τώρα. υπέ Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 17 υπέ Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 18 υπέ Κατά αποχές. απορρίψεται. Αλλά θέλει έλεγχο. Η 18 παρακαλώ ξανά. Αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 ε, και 26 ειπε Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική d υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είμαστε στην 45 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη 46. Παρακαλώ ψηφίστε. Και αν ψηφίσατε όλοι κλείνει. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική σε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές απορρίψεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55. Όχι, η συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική γιώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική μη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και που πάμε τώρα στην 82 ψήφι υπέρ κατά αυτό θέλει έλεγχο παρακαλώ την τροπολογία 82 αρχίζει τώρα ο έλεγχος ψηφίσατε όλοι πέρας Απορρίπτεται. Συμβαστική κάπα υπέ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 102 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική N υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ομικρόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική π υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έχει 113 υπέρ. Κατά. Αποχές Έλεγχο στην 113. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίψετε. Με μικρή διαφορά πλην απορρίπτεται. 114 υπέρ κατά αυτό θέλει και αυτό έλεγχο 114 ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά. Δεν καταλαβαίνω τι ψηφίζετε. Λοιπόν, 116 ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ε, με μια ψηφοδιαφορά πάλι. Απορρίπτεται. Συμβαστική ΕΡ υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Η 118, 20 συγγνώμη, υπέρ κατά 120 απόχες. Και αυτό θέλει έλεγχο. Η τροπολογία 120, ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. φέρες Και με μικρή διαφορά απορρίπτεται. Ωραία. Συνολική τώρα, τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία για όλη την έκθεση. Αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται η έκθεση. Α, έπρεπε να είχα ψηφίσει κι εγώ. Μα δεν μου λέτε τίποτα εδώ πέρα. Τώρα πρέπει να ψηφίζω κι εγώ. <laughs> Το προηγούμενο όχι. Λοιπόν, άμα με αφήνετε παίζω κι εγώ, άρα πρέπει να μου το λέτε. Λοιπόν, πέρα της ψηφοφορίας, αποτέλεσμα 38 υπέρ, 9 κατά και 8 αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Συγκητρία. Ε, τι Παρακαλώ, εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και ιδίως τους κοιόδης εισηγητές, καθώς επίσης και όλους τους συνεργάτες οι οποίοι πραγματικά μας επέτρεψαν να συντάξουμε και να υπερψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα τον κατάλογο της ψηφοφορίας ε, για να φτάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Ε, έχουμε πολλές τροπολογίες, 44 συμβαστικές, τέσσερις ε, συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών. Πολύ δουλειά λοιπόν έχει γίνει, κάτι που φαίνεται και από τον όγκο του καταλόγου ψηφοφορίας. Να λοιπόν στην πρώτη τροπολογία, τροπολογία 87 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 96 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται και οι 105 είναι ταυτόσιμες. Ψήφισαμε δηλαδή και τις δύο μαζί. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά. Να το ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 115 αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Έχουμε έναν παραπάνω από τους σοσιαλδημοκράτες. Ε, Γιούτα, για μέτρησε τα πρόβατά σου, σε παρακαλώ. 115, ωραία. Εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε καλύτερα. Η ηλεκτρονικός έλεγχος 124. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Να την ελέγξουμε. 128 ηλεκτρονικός έλεγχος. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. 130 ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ε, συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 169 κατά τμήματα σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. ΦΕΜ 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φεμ. Φεμ 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την ελέγξουμε. 174. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται σαφώς 175 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΦΕΜ 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 187 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 188 ε, είναι ταυτόσημη. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΕΜ 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και οι 195 είναι ταυτόσιμες. 200 και 201 είναι επίσης ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ήθελα να το ελέγξουμε. 200 και 201 ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 27-27. 205 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 198 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 202 και 203 υπέρ, κατά, να το ελέγξουμε. 202-203. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Λήξη τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 204 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να το ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηλά το χέρι, διότι τελειώς δεν βλέπουμε. Ε, ψηφίσατε όλοι, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 17. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Φεμ 3. Μόνο το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 226 και 227 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συμβαστική 20 υπέρ, κατά, Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 239 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24. Σωστά. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 248 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΕΜ 25. Καταπίπτει, ε? 251 υπέρ κατά αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ, τη 251 ηλεκτρονικός έλεγχος. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 253. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 257 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΦΕΜ 28. Ψηφίζουμε. ΦΕΜ 28. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΕΜ 6. συμπεριλαμβάνεται χωρίς ψηφοφορία. Ε, συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΕΜ 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 277 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Συμβαστική 33 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Απορρίπτεται. ΦΕΜ 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτήν θα ήθελα να την ελέγξουμε. ΦΕΜ 16. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 34. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 284 με μια προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μικρή διαφορά. Ε, η άλλη έχει αποσυρθεί. Συμβαστική 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 290 παράδεκτη. 293. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 294 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 301. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 311. Ε, καταπίπτει 308 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 312 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική, μάλλον όχι, να την ελέγξουμε, την 312. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ, λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 314 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 316 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε 316 ψηφίσατε παρακαλώ όλοι λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται 318 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 320 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το ίδιο ισχύει για την 321. Είναι ταυτόσημη μάλλον. 322 υπέρ.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 Οι 320 και οι 321 εγκρίθηκαν, άρα καταπίπτει η 322. Ωραία, 323 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 325 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 328 υπέρ κατά για να δούμε, να ελέγξουμε. 328. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 329. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 330. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε πάλι. 330. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 331 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 332 υπέρ. 332 υπέρ. Εγκρίνεται μάλλον. 333 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος της 333. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 334 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε πάλι την 334. ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 337 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 339 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 340 και 341 και 342 είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά. Να το ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Εγκρίνεται. Φτάνουμε στην 347 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. 347 ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 349 υπέρ. Κατά. Είναι σαφές. Απορρίπτεται. 350. Καταπίπτει. 351 καταπίπτει. Τριακόσια υπέρ, κατά, να το ελέγξουμε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Απορρίψετε με μικρή διαφορά. «353 υπέρ». Κατά. Να το ελέγξουμε και αυτό. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Σαφές είναι το αποτέλεσμα, εγκρίνεται. 355 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε και αυτήν. Ζήτω συγγνώμη, λάθος του σκηνοθέτη. Καταπίπτει. 356 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 360 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 300 και 310 υπέρ κατά να το ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Das Απορρίπτεται. Συμβαστική 43 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Συμβαστική 43. Ελέγχουμε. Alle abgestimmt, dann schließen wir. Das ist ab. Απορρίπτεται. Ε, 358 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 267, Amendment 267 dafür. 267 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την ελέγξουμε. 267 ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Και φτάνουμε στην 359 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φεμ 8. Όχι. Φεμ 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φεμ 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φεμ 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά. Θα ήθελα να την ελέγξουμε. Την ΦΕΜ 14, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. ΦΕΜ 17 συμπεριλαμβάνεται χωρίς ψηφοφορία. ΦΕΜ 20 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Φέμ 21 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Φέμ 22 υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την ΦΕΜ 22, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται, σαφώς. Θέμη 23. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 24 δεν ψηφίζουμε. Θέμη 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θέμη 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΕΜ 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τηλέφωνο 370 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 371 προτείνεται να ψηφίσουμε μαζί τις τροπολογίες από 371 έως 382. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Πάρα πολύ ωραία. Υπέρ. Όχι. Έχουμε αντίρρηση. Ωραία. Θα τους ψηφίσουμε μία-μία. 371. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 372 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 373 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 374 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 375 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 376 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 377 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 378 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 379 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 380 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 381 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 382 υπέρ κατά κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία. Φτάνουμε λοιπόν τώρα στην 44, ε, συμβαστική 44 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 385 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ,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 και 21 μαζί είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές να την ελέγξουμε την 30 ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίσατε παρακαλώ όλοι κλείνουμε την ψηφοφορία εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά δύσκολο. 31 να την ελέγξουμε. Haben alle abgestimmt. Dann ist die Abstimmung geschlossen. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σας παρακαλώ, ε, αν σηκώνετε πιο ψηλά το χέρι θα είναι λίγο πιο εύκολο για μένα. 32. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Φεμ H. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 36 αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 38. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σαράντα εννέα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πενήντα με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά θα ήθελα να το ελέγξουμε ελέγχουμε την 53 ηλεκτρονικά ψηφίσατε παρακαλώ όλοι λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται 54 υπέρ κατά Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Φεμ α, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φεμ β. Δεν την ψηφίζουμε. σι, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. 56 διορθώνει ο πρόεδρος. 56 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά αποχε... απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε παρακαλώ την 59. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές Σας παρακαλώ να την ελέγξουμε. Τροπολογία 61, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 62, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64, υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. 64, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Ναι. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε επίσης την 65. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Ωραία. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές θα παρακαλούσα να την ελέγξουμε νομίζω ότι απορρίπτεται 67 ψηφίσατε παρακαλώ όλοι ναι και πράγματι απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 καταπίπτει. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 μέχρι 86 όλες μαζί αν δεν υπάρχει αντίρρηση. Υπάρχει αντίρρηση? Καμία αντίρρηση. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε είσαι υπεύθυνο για, την υγεία εδώ στην Επιτροπή, έτσι δεν είναι. Ε, ωραία. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να την ελέγξουμε θέλετε. 81, να την ελέγξουμε. Das ist angenommen. Εγκρίνεται. Ε, 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φεμ ή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φεμ G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φεμ I υπέρ κατά υπέρ κατά να την ελέγξουμε. Φεμ I ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Ναι, ωραία εγκρίνεται FEMJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται FEMK υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται FEML υπέρ κατά να την ελέγξουμε FEML ελέγχουμε ηλεκτρονικά ψηφίσατε παρακαλώ όλοι ναι ισοψηφία απορρίπτεται FEMM υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά ΦΕΜ, M ψήφισατε παρακαλώ όλοι από ό,τι φαίνεται ναι απορρίπτεται Φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία για το σύνολο της έκθεσης. Σε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Από τους συναδέλφους μου ποιος θα αποσυρθεί. Γιατί εγώ δεν αποσύρωμαι, θα ψηφίσω. Τώρα εντάξει, γιατί ήμασταν ένα υπεράριθμος από την Λοιπόν, αποτέλεσμα 44 υπέρ, 9 κατά, με μία αποχή. Υποθέτω ότι συμφωνείτε να προσθεθεί ονομαστική ψηφοφορία στην έκθεση. Ήθιστε και στην προηγούμενη έτσι κι αλλιώς, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι έχουμε εδώ. Έχουμε μια κάπως μικρότερη γνωμοδότηση. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt. Πάμε στο σημείο 8 λοιπόν. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 3 υπέρ. Τι έγινε, καταπίπτει αυτή. Ωραία. Η 4 υπέρ. Κατά. Λάθος, διορθώνει ο πρόεδρο. Λοιπόν, ε, γινάμε πίσω λίγο γιατί κάναμε ένα λάθος. Η τροπολογία 3. Πρέπει να ψηφιστεί. Ψηφίζουμε την 3. Υπέρ. Κατά. Για να το ελέγξουμε αμέσω. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίψετε. Η τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές σύμβαση Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 12 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική β. Τσεκ, φωνές από κάτω. Ωραία, ας το ελέγξουμε. Την τροπολογία 12, έτσι, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική βήτα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται η τροπολογία 19 σε τμήματα είναι αυτή. Τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική σε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 24 και πάλι κατά τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, άκουσα πάλι τσεκ Είπε κανείς, ωραία, να την ελέγξουμε. 37, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψήφισατε όλοι, πέρας. Μμμ, απερίφθη. Η 37. 38, έχει διεκπαιρεωθεί μάλλον, έτσι. 39, Είπε κατά. Α, αυτό θέλει έλεγχο. Η 39, παρακαλώ, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Mm. Ισοψηφία. Απορρίψετε. Η 40 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίψετε. Η 43 χωριστή ψηφοφορία τρίμα πρώτο υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται η δεύτερη υπέρ. Το δεύτερο τμήμα κατά και αυτό θέλει έλεγχο. Το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 43. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42 υπέ Κατά. Και αυτό θέλει έλεγχο και πάλι. Η 42 η ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Περές. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. Η 45 υπέρ. Κατά αποχές. Ε, απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές. Αυτό θέλει έλεγχο. Η 46 συγκεκριμένα ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. Η 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 47 έλεγχο θέλετε, ας το ελέγξουμε λοιπόν. 47 ηλεκτρονική επαλήθευση.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 Συγγνώμη, δεν είχατε ψηφίσει όλοι, το κλείσαμε νωρί. Επαναλαμβάνεται η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 57. Έτσι όταν είσαι πολύ βιαστικός συμβαίνουν και τέτοια. Αγκρίθηκε τώρα. Η 57. Και να μην μας κατηγορήσει κανείς ότι δεν αφήνουμε την ψηφοφορία και την κλείνουμε πολύ νωρίς πριν υπάρξει αποτέλεσμα. Λοιπόν, 58 υπέρ κατά έλεγχος πάλι για την 58 ηλεκτρονικά. Haben Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε συμβαστική F κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική H κατά αποχές εγκρίνεται η 64 έχει αποσυρθεί και πάμε στην 65 κατά τμήματα τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ερχόμαστε στο σύνολο της ψηφοφορίας για όλη τη γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Ε, Ένα υπεράριθμο από την ΚΟΕ, βγάλω τη δική μου κάρτα για αλλαγή. 44-10, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ωραία. Και πάλι θα το ε, επισυνάψουμε το αποτέλεσμα της ονομαστικής ψηφοφορίας ως ήθιστη στην έκθεση. Πάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία μας που είναι το σημείο 9 η κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και τα λοιπά και ανάγκη η τροπολογία 1 ψήφι υπέ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική α υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 10. Η 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 11 υπέρ κατά έλεγχος παρακαλώ. Ηλεκτρονικά ελέγχουμε την 11 τροπολογία. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται σαφώς. Μετά έχουμε, ποια τροπολογία έχουμε, τη 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται συμβαστική β υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική σε υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική G υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 44 τώρα υπέρ κατά. Τι έγινε, τη 44 ψηφίζουμε το. 44. Το είπα και 44. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ για τη 44. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίψετε. Η 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 46 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε. Η συμβαστική έτσι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 54 με μια προφορική εδώ τροπολογία που βλέπετε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά έλεγχος παρακαλώ ηλεκτρονικός για την τροπολογία 56. Ψηφίσατε όλοι. Yes. Έτσι φαίνεται. Απορρίψετε. 57 υπέρ κατά αποχές. Απορρίψετε. Συμβαστική γιώτα υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές. Απορρίψετε. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική και υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολόγια 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ τσεκ απερίφθη, λάθος το έκανα. Εγώ φταίω. Τυπογραφικό λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα θέλετε έλεγχο για την 79. Ε, εγώ, εμείς δεν είμαστε τόσο... Ε, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε 80 είπε, Κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 85 με μια ε, προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 υπέρ όχι είναι ταυτόσιμη με την 90 μαζί λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται η συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έχουμε την 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 δεν ψηφίζεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά το θέλει έλεγχο, η 97 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίψετε, 20-30, 98 υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. Το σύνολο τώρα του σχεδίου γνωμοδότησης. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Εψηφίσατε όλοι. Ωραία καλησπερα 42 42-9. Συγχαρητήρια στην κυρία Μωρέν Σαχτιέ. Ελίζαμπετ. Ελίζαμπετ. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ή τουλάχιστον αυτό ελπίζω. Με τις ψηφοφορίες. Καλό σας ε, μεσημερινό διάλειμμα που είναι λίγο μεγαλύτερο. Ραντεβού στις 3. Oh.